δουλειά μας είναι να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων. Οι αποκαλύψεις οι σχετικές με την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εκπλήξει. Βέβαια στην κατασκοπία αποδίδει το στοιχείο της έκπληξης, του ευνηδιασμού. Βέβαια Κανείς προσδοκά, περιμένει το να τον κατασκοπεύει κάποιος άλλος. Οπότε γι' αυτό και εμείς είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας. Αυτό που μας εξέλιξε ήταν ε, το βελνικές των ικανοτήτων αυτών που μας παρακολουθούσαν. Εμείς έχουμε επαρκή προστασία και πλαίσιο ασφάλειας. Όλα αυτά είναι αριθμισμένα και αποπτεύονται. πιο πολλοί αυτοί που μας εποπτεύουν παρά αυτοί που δουλεύουν για την Europol, ξέρετε. Αυτά, επομένως, διαπνέουν όλη την ε, διαδρομή κάποιου που δουλεύει εκεί και υπάρχουν έλεγχοι σε πολλά επίπεδα, παρακολούθηση συστημάτων κλπ. Μας ε, εποπτεύει η Επιτροπή Ασφαλείας της Europol. Πρόκειται για εμπειρογνώμες από τα κράτη-μέλη. και συμβουλευόμαστε αυτή την Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Κάθε καινούριο σύστημα, κάθε αλλαγή στα συστήματα που έχουμε περνάει από αυτή την Επιτροπή για να εγκριθεί, για να πιστοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Μπορούν να πιάσουν δουλειά στην Europol μόνο πρόσωπα που έχουν την ηθαγένεια κάποιες χώρες της και που έχουν περάσει από έλεγχο από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Έχουμε βέβαια κάποια τροτά σημεία. Έχουμε εξωτερική κυκλοφορία δεδομένων και εξαρτώμεθα και από κάποια κέντρα πληροφορικής, κάποιες υπηρεσίες που είναι εξωτερικά. Βέβαια έχουμε κάποιο είδους υπεργολαβίες που γίνονται και αφορούν όμως μη επιχειρησιακά συστήματα. Όλοι οι σύμβουλοι που συνεργάζονται μαζί μας για τα θέματα ε, πληροφορικής, θα πρέπει να ελεγχθούν από ασφαλείας ε, εκ των προτέρων. Και η δουλειά τους εποπτεύεται από, από τα μέλη της Europol. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα τα οποία αφορούν τον επιχειρησιακό μας κλάδος και επίσης δεν χρησιμοποιούμε το σύννεφο, το cloud, ε, ούτε κάποιο είδους τρόπους εξωτερικής φιλοξενίας και απο, ή αποθήκευσης όσον αφορά τις υπηρεσίες τις ε, επιχειρησιακές. Οπότε τώρα όσον αφορά τα δεδομένα συνεργαζόμαστε με εθνικές ε, υπηρεσίες και υπάρχει κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων που κυκλοφορούν στο δίκτυο firewalls πριν από οποιαδήποτε συνεργασία και μεταφορά δεδομένων προς τρίτη χώρα. δεν έχουν πρόσβαση και δεν, δεν, δεν είναι ορατά τα δεδομένα της Europol από άλλες υπηρεσίες ή από διοικητικές αρχές κρατών μελών συμμετέχουμε στην υπηρεσία ε, ανταλλαγή πληροφοριών υποστασία δομένων και στο ΛΙΣΑ. Γενικά θεωρούμε ότι οι υπόλοιπε υπηρεσίες τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεν έχουν τόσο αυστηρή, ε, αυστηρούς κανόνες ασφαλείας όπως εμείς. Και επίσης το προσωπικό μας προέρχεται από τις διοικητικές αρχές και είναι εξοικειωμένοι λοιπόν με τέτοιου είδους ε, πλαίσια και κανόνες προστασίας δεδομένων. Επίσης, Και έχουμε και κάποια τροτά σημεία, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν να κάνουν με την φύση που λειτουργούν κάποια θεσμικά όργανα που έχουν λιγότερη ασφάλεια από ότι εμείς. Το αυτό αφορά και την αποθήκευση δεδομένων στο, στο νέφος, στο σύννεφο, στο cloud. Επίσης υπάρχει έκθεση στο διαδίκτυο των συστημάτων πυρήνα του ΚΟΡ. Επίσης άλλα δυνατά σημεία είναι κάποιες, ε, κάποια gadgets τα οποία είναι, ανήκουν σε κάποια πρόσωπα που δουλεύουν στην υπηρεσία, ε, το, στο ασύρματο δίκτυο, ε, όπως επίσης και, και τα ε, κυκλοφορία δεδομένων στο ίντερνετ. Θα πρέπει με τη δουλειά μας να δείξουμε στους εταίρους μας τι έγινε ε, και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να προστατευτούμε ε, για το πώς δεν θα έχουμε τέτοιου είδου ακούσια, κατασκόπευση και υποκλοπή δεδομένων. Αυτά κύριε Πρόεδρε και περιμένω τις ερωτήσεις της τυχόν και πρόθυμα να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Τήρησατε τα χρονικά όρια. Όμως, δεν μιλήσατε, δεν εξαντλήσατε όλο τον χρόνο, από ευθύ αμέσω πάντω να προχωρήσουμε στον δεύτερο συγγνώμη, τον κύριο Ούντο Χέλμπερ, που είναι εκτελεστικό διευθυντή τη ΕΝΗΣΑ και εσεί κύριε έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο. Μια αρχική παρατήρηση. Η βασική μας δουλειά στην Μίζα είναι να εξετάζουμε τις νέες τεχνολογίες, ε, επιχειρηματικά μοντέλα και ασφάλειες ε, και ε, απειλές, με συγχωρείτε, τις ασφάλειες των υπολογιστών. Εάν μιλήσουμε λοιπόν για τη μαζική αυτή παρακολούθηση, θα ήθελα να πω πως η ΕΝΙΖΑ, η εντολή της ΕΝΙΖΑ δεν συμπεριλαμβάνει την κατασκοπία. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι μπορώ να συνεισφέρω στη συζήτηση. Θα ήθελα να μπω, θα ήθελα να εστιαστώ στο θέμα της ιδιωτικής ζωής. Ένα από τα δύο βασικά ζητήματα της ασφάλειας ε, εδώ πέρα είναι η εμπιστευτικότητα και η ακαιρεότητα, δηλαδή είτε να μην χάνονται και υποκλέπτονται τα δεδομένα, είτε να μην τα αλλάζουν κιόλας να σας δώσω κάποια παραδείγματα και συστάσεις. Εάν δείτε τη σημερινή συζήτηση, μιλάμε για προστασία προσωπικών δεδομένων, διατήρηση δεδομένων, έχουμε διαφορετικά συμφέροντα εδώ πέρα. Επίσης, αν δείτε την Ευρώπη, υπάρχει διαφορετική αντίληψη της ιδιωτικής ζωής από τις είπα και το μήνυμά μου βεβαίως ε, είναι αυτό με τα κόκκινα γράμματα. Δηλαδή, στα σημερινά επιχειρηματικά μοντέλα πλέον ε, το νόμισμα είναι τα προσωπικά δεδομένα ή αλλιώς σε κάποιες περιπτώσεις ο νόμος μπορεί να καταστρέψει επιχειρηματικά μοντέλα εταιριών μεγάλων που προσφέρουν υπηρεσίες ε, στο νέφος το λεγόμενο. Μια άλλη σημαντική εμπειρία που έχουμε είναι μια μελέτη που κάναμε στη Γερμανία όπου υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτική ζωή. Απ' τη μία λένε είναι σημαντική ασφάλεια της πληροφορικής, αλλά από την άλλη υπήρξε μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο που προσφέρουμε κάποια εισιτήρια και τους λέμε αν θα μας δώσετε το νούμερό σας για 50 cents λιγότερα, το νούμερο του τηλεφώνου. Και βλέπετε 87% τις 100 των χρηστών έδωσαν το νούμερό τους του τηλεφώνου για 50 cents. 50 ε, λεπτά του ευρώ. Βλέπετε λοιπόν πως λέγεται εδώ πέρα πως ο καθένας ε, έχει το δικαίωμα στην ε, προστασία των δεδομένων. Έχουμε το οδηγία του 1995. Βεβαίω συζητάμε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή από διαφορετική σκοπιά και όταν έχουμε νέες τεχνολογίες, εάν δείτε την ιστορία, όταν οι νέες τεχνολογίες γίνονται επιχειρηματικά μοντέλα, τότε ε, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αν δείτε τα δεδομένα, ε, μπορούμε να σας δείξουμε τον κύκλο ζωής των δεδομένων. Συλλέγονται τα δεδομένα, τα χρησιμοποιεί κανείς, ε, τα συσχετίζει με άλλα δεδομένα, τα αποθηκεύει, τα ανακτά και μπορεί στο τέλος, ανάλογα με το μοντέλο, να διαγραφούν. Και Βεβαίως ε, μιλάμε για διαφορετικά σημεία στην ζωή των δεδομένων και αν μιλάμε για κεραιότητα ε, και λοιπά χαρακτηριστικά των δεδομένων, μιλάμε για διάφορα, διαφορετικά σημεία του επιχειρηματικού μοντέλου. Εδώ πέρα βλέπετε τα δεδομένα τα σημερινά στο διαδίκτυο και το πώς πρέπει να τα προστατεύσουμε. Έχουμε δεδομένα που μοιράζονται στον κόσμο. Αν δείτε το Google+, Plus, δεν το χρησιμοποιούμε πολύ αυτή τη στιγμή. Εάν δεν θέλετε να τα εκθέσετε, μπορείτε να μην τα βγάλετε στο ίντερνετ. Αλλά αλλά όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα ε, βλέπετε ότι αφορούν αμερικανικές εταιρείες, έτσι. Μετά, έχουμε πολλές ε, παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Αυτά εδώ είναι από τα τελευταία χρόνια τα συμβάντα. Πάνω από 30.000 ε, αρχεία εκλάπησαν. Θα θυμάστε πριν από κάτι χρόνια η Sony έχασε τα δεδομένα των χρηστών του PlayStation Network και άλλες εταιρείε ε, μπορεί να μην ξέρετε καν πού αποθηκεύονται τα δεδομένα σας. Αυτό είναι από το γραφείο της ε, Κομισιόν ε, παραβιάσει συστημάτων δεδομένων. Και νομίζω είναι ενδιαφέρον να δείτε τον κανονισμό για την ειδοποίηση της παραβίασης του δικτύου δεδομένων ε, για να μπορέσετε να συγκρίνετε γιατί αν έχετε μία τέτοια παραβίαση καμιά φορά δεν είναι υποχρεωτικό να το δηλώνει κανείς και βεβαίως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν έχει κανείς στατιστικά στοιχεία. Βεβαίως Αυτό είναι εδώ πέρα κάτι το οποίο κάναμε μαζί με την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Ξεκινήσαμε το 2012 και το 2013 το οριστικοποιήσαμε με την τεχνική υποομάδα. Το νόημα είναι λοιπόν να δώσουμε περισσότερη προστασία όταν ε, έχουμε δεδομένα και βεβαίως προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και τις τεχνικές ικανότητες της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Αυτό θα δημοσιευτεί σε λίγες μέρες. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες δηλώσεις για την κρυπτογραφία και το δικαίωμα το λεγόμενο να ξεχαστεί κανείς που δεν συζητάμε. Το μήνυμα εδώ είναι το εξής. Αν μιλάμε για προστασία δεδομένων, τότε έχουμε πολλές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλά δεν χρησιμοποιούνται, δεν εφαρμόζονται ή δεν συμφέρουν, ε, δεν αποδίδουν οικονομικά για τις εταιρείες. Τι εννοώ δηλαδή, υπάρχει κρυπτογράφηση, διαφορετική τύπη κρυπτογράφησης, πολύ δύσκολη να σπάσει και πρέπει να το σκεφτείτε ε, στην ιδιωτική σας ζωή. Το θέμα όμως είναι πόσο καιρό πρέπει να είναι ασφαλή τα δεδομένα για σας ή την επιχείρησή σας. Εάν υπάρχει ένα έργο για, για έξι μήνες και μετά δεν χρειάζεστε παραπάνω τα δεδομένα αυτά, αν έχετε παραδείγματο χάρη, αν έχει η εταιρεία σας ή εσείς εδώ πέρα, αν έχετε μια συνάντηση με μια εκπροσώπηση ενός άλλου κράτους και κλεισμένων των θυρών, ε, σε μερικές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κρατάτε τα δεδομένα πάνω από κάνα δύο μέρες. Οπότε αρκεί να είναι δύσκολη η αποκρυπτογράφηση και η πρόσβαση, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να είναι ασφαλή τα δεδομένα για χρόνια ή δεκαετίες. Ε, τότε χρειάζεται πολύ ισχυρότερη κρυπτογράφηση, αλλά υπάρχουν πολλές διαθέσιμες τεχνολογίες. Το ίδιο επίσης για ηλεκτρονικές υπογραφές. Υπάρχει αυτή η τεχνολογία εδώ και 10 χρόνια. Αλλά εξακολουθούμε να στέλνουμε email τα οποία ε, είναι σαν κάρτ ποστάλ, έτσι. Όλοι το διαβάζουν και όλοι μπορούν να το αλλάξουν. Οπότε με τις τεχνολογίες αυτές μπορούμε να έχουμε ασφαλή email. Μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν αυτά, αλλά το μήνυμα είναι το έχουμε και ε, φέτος για πρώτη φορά βγάλαμε μια σύσταση από την ΕΝΙΖΑ για αυτά τα θέματα γιατί ε, υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις σε εθνικές γλώσσες των κρατών μελών αλλά προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιες δημοσιεύσεις τουλάχιστον στα αγγλικά σε όλες τις χώρες οπότε τα βασικά μηνύματα όπως είπα είναι πως η τεχνολογία υπάρχει Απλά να φτάσω στο συμπέρασμα. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Είμαστε σε θέση να γνωμοδοτήσουμε. Επίσης ε, στηρίζουμε το ότι η οδηγία πρέπει να προωθήσει την ειδοποίηση και άλλων κλάδων και πρέπει να υπάρχουν ε, σχέσεις με την πολιτική και τις ερευνητικές πρωτοβουλίες. Εδώ πέρα έχουμε μια διαφήμιση με την επόμενη ελληνική προεδρία. Στην Αθήνα 20-21 Μαΐου του 2014. Σας ευχαριστώ Ούντο, κύριε καθηγητά. Τώρα περνάμε στο τρίτο μέρος, μέλος με συγχωρείτε, του πάνελ, τον κύριο Φλόριαν Βάλτερ. Σύμβουλο για θέματα πληροφορικής και επικοινωνίας και τεχνολογίας για τα επόμενα για τα επόμενα 10 λεπτά. Γεια σας, λέγομαι Φλόριαν Βάλτερ, είμαι Γερμανός και τα τελευταία 12 χρόνια εργαζόμουν ως σύμβουλος ασφάλειας και δοκιμαστής ασφάλειας. Έχω Δύση σε ένα σωρό συστήματα. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Με ε, συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με δίκτυα ολόκληρα, με οχήματα, οτιδήποτε διαθέτει ένα IP, ένα πρωτόκολλο τέλο πάντων και ένα σύστημα πληροφορικής. Δεν έχω φέρει καμία παρουσίαση μαζί μου, αλλά έχω κάποιες καλές συμβουλές μετά από δεκαετή εμπειρία. Το πρώτο που θα πρέπει να καταλάβετε είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια και ποτέ δεν θα υπάρξει. Η ασφάλεια είναι πάντοτε κάτι που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Πρέπει να ε, ε, ε, ισοζυγιάζει κανείς τα πράγματα. Δεν μπορεί στην ασφάλεια να είναι κανείς 100% ασφαλής. Πρέπει κάποια πράγματα απλώς να εξοβαλίζονται. Είναι εξισορρόπηση μεταξύ της χρήσης και της ασφάλειας. Εξισορρόπηση μεταξύ κόστους και ασφάλειας. Δεν μπορεί να έχει κανείς απόλυτη ασφάλεια 100%. Μπορεί απλώς να βάζει τον πύχη ψηλά. Τόσο ψηλά όσο χρειάζεται να βάζει σε δύσκολη θέση τους hackers, να μην μπορούν να σας παραβιάσουν το δίκτυο και να το, ε, να, το, να δυσδύσουν σε αυτό και να αποσπάσουν στοιχεία από αυτό επίσης. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νόμους που δίνουν τη δυνατότητα σε ενώσεις οργανώσεις και κυβερνητικούς φορείς να αποκρύψουν πληροφορίες περί προβλημάτων ασφαλείας και ευάλωτα σημεία του, συστήματό του συστήματός τους καθώς οι εταιρείες, φορείς, οργανώσεις, ενώσεις και κυβερνητικοί φορείς μπορούν να αποκρίνουν τις πληροφορίες που ήδη διαθέτουν για προβλήματα ασφαλείας σε κοινά συστήματα πληροφορικής δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κανείς να τα καταφέρει. Διότι τα ξέρουν με τα παραθυράκια, ενώ εσείς δεν τα ξέρετε. Πώς να υπερασπιστεί κανείς τον εαυτό του ε, απέναντι σε παραθυράκια τα οποία δεν γνωρίζει καν, τον οποίο αγνοεί την ύπαρξή τους. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι του προβλήματος. Τέτοιοι νόμοι εγκρίθηκαν μέχρι και εδώ. Ήμουν στην συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για να καταψηφίσω. Κανείς δεν με άκουσε. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να δείτε είναι ο προπολογισμό. Η ε, ΕΝΙΣΑ έχει προπολογισμό η NSA έχει προπολογισμό 56 δολάρια ετησίω. Πόσο είναι ο προπολογισμό σα για την ασφάλεια πληροφορική και πόσο είναι ο προπολογισμό σα για το ε, χαρτί υγείας. Μάλλον είναι υψηλότερο. Για σκεφτείτε το. Και επίσης δεν μπορεί να θεωρείτε ότι δεν θα δεχτείτε επίθεση, ότι δεν θα σας κάνουν hacking αν δαπανείτε περισσότερα, δαπανάτε περισσότερα για, την, για το χαρτί υγείας από ότι για την ασφάλεια στο ίντερνετ η NSA έχει ακόμη περισσότερα κονδύλια από όλου τους ευρωπαϊκούς θεσμούς συνολικά αν έχουν καν ασφάλεια IT. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο προπολογισμού, είναι και θέμα γνώσης του προσωπικού και των εργαζομένων σας. Πόσο σίγουροι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στο τμήμα IT, πόσο καλά καταλαβαίνουν τα συστήματα που ε, πρέπει να φροντίσουν. Ξέρετε τι κάνουν. Μάλλον όχι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάλλον και αυτοί περιορισμένες γνώσεις για τα συστήματα που χρησιμοποιούν. αγοράζουν έτοιμο ε, ε, από αμερικανικές εταιρείες κατασκευασμένο λογισμικό. Οι εταιρείες εκείνες έχουν τα δικά του συστήματα ασφαλείας. Ίσως να έχουν φτιαχτεί, να έχουν ε, δεχτεί την επίδραση της NSA. Πώς θα είναι το σύστημά σας ασφαλές εάν ξεκινάτε ήδη με τέτοια λειτουργικά, με λογισμικά που είναι κατασκευασμένα από άλλους. Το έχετε σκεφτεί ποτέ. Για σκεφτείτε το. Θα έπρεπε. Ως ε, επιτιθέμενος έχει κανείς ένα στρατηγικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με αυτούς που πρέπει να υπεραμεινθούν των συστημάτων τους. Ως επιτιθέμενος πρέπει κανείς να βρει απλώς μία ε, κερκόπορτα, μία χαραμάδα, μία δίωδο. Ενώ αυτός που υπερασπίζεται το σύστημα πρέπει να τις βρει όλες και να τις καλύψει. Πρέπει λοιπόν κανείς να έχει πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και αρκετούς πόρους, αλλά και καλά συστήματα για να προστατέψει τις δομές του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα και την ικανότητα να συνειδητοποιήσει, να αντιληφθεί πότε πέφτει θύμα επίθεσης. Για τους hackers υπάρχουν δύο οργανώσεις στο διαδίκτυο. Αυτές που ξέρουν ότι μπορούν να δεχτούν επίθεση και ότι δέχονται και αυτοί που δεν το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι μάλλον στη δεύτερη ομάδα. Για σκεφτείτε το και αυτό. Χρειάζεστε άμεση αντίδραση στα περιστατικά. Πρέπει να μπορείτε να αντιμετωπίζετε τις επιθέσεις μόλις συμβαίνουν, όχι έξι μήνες μετά. Γιατί θυμηθείτε, οι καλύτεροι επιτιθέμενοι, οι πιο αποτελεσματικοί, είναι αυτοί που δεν τους ανακαλύπτει καν κανείς. Και αυτοί οι hackers, αυτοί ειδικά που χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις, είναι ου, πολύ καλοί. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και ξέρουν να έξω και ανακατατά τα συστήματά σας και το προσωπικό σας. Καλύτερα και από ό,τι οι εργαζόμενοι εδώ. Όταν ένας επιτιθέμενος επιτίθεται σε από τα συστήματά σας, έχει το πλεονέκτημα. Σας είπα, πρέπει να βρει μία τρύπα. Μία δίωδο για να μπει στο σύστημά σας. Με το που θα μπει όμως, με το που θα μπει στο σύστημά σας, αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα μετατοπίζεται και περνάει στα χέρια του ε, ε, αμυνόμενου. Διότι εσείς γνωρίζετε και χειρίζεστε το σύστημα. Εσείς γνωρίζετε το υλικό που χρησιμοποιείτε. Αλλά πρέπει πρώτα να το αντιληφθείτε για να τους πιάσετε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεστε πολύ καλή και εγκαιρή απόκριση στα περιστατικά. Πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητε να αντιληφθείτε καταρχά πότε δέχεστε επίθεση. Οι περισσότεροι από εσά τώρα θα σκέφτεστε το λογισμικό κατά των ιών, τα ε, συστήματα πρόληψη των ε, ε, παραβιάσεων ή τη αντιμετώπιση των παραβιάσεων. Αυτά μπορείτε να τα αγοράσετε και έτοιμα πολλέ φορέ από την Αμερική με υψηλότερε τιμέ. Να σα πω κάτι, Συνήθω είναι ήδη πειραγμένα. Μην σκέφτεστε τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν τέτοια λογισμικά ασφάλειας που ουσιαστικά να αφήνουν και άλλα διόδους ανοιχτές στο σύστημα ασφάλειας σας. Η... Ο συνδυασμό δεδομένων είναι κάτι από τα δυσκολότερα πράγματα που μπορεί να κάνουν οι προγραμματιστές. Έχετε ουσιαστικά πολλαπλασιάσει επί χίλια το σύστημα της το τα σημεία του συστήματος ασφάλειας, εάν τα χρησιμοποιήσετε. Αυτοί όμως που προσέχουν το σύστημά σας, εάν είναι καλά εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι και γνωρίζουν καλά το σύστημα, τα γνωρίζουν απ' έξω και ανακατοτά, τότε μπορεί και να αντιληφθούν ότι κάτι πάει στραβά, εάν κάποιος ε, μπει στο σύστημα και πειράξει ζωτικές λειτουργίες του συστήματος προκειμένου να επωφεληθεί ως επιτιθέμενος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να έχει έναν administrator, ένα χειριστή που να ασχολείται με χιλιάδες πλευρές του συστήματος. Αν το σύστημα είναι μεγάλο, πρέπει να έχει έναν που θα γνωρίζει όλο το σύστημα. Για να συνοψίσω, η περιπλοκότητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της ασφάλειας. Να το θυμάστε, μόλις ζητάτε ένα καινούριο χαρακτηριστικό από το τμήμα IT σας να έχετε καλύτερες και περισσότερες ε, δυνατότητες και πόρους. Χρειάζεστε μάλλον περισσότερους εργαζομένους και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι και να γνωρίζουν τα συστήματά τους πολύ καλά. Επί της ουσίας, αυτά είχα να σας πω συμβουλές για να έχετε καλύτερη ασφάλεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βόλτερ ανεξάρτητος σύμβουλος πληροφορικής και τεχνολογίας. Ε, να σας πω, επειδή το αναφέρατε, να σας πω ότι θερμά εκτιμούμε τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων μας στο πάνελ και στην Επιτροπή μας, ιδιαίτερως τι δικές σας, απλώς να σας βεβαιώσω, όταν όπως τόσοι άλλοι προσκεκλημένοι ε, παρεμβαίνετε και μας μιλάτε, κάποια από εμάς ακούμε. Σας ακούμε πραγματικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και για άλλους λόγους, όχι μόνο γι' αυτό. Για να σκεφτούμε, να κρίνουμε και να διαμορφώσουμε δική μας ε, γνώμη και να χειριστούμε το χρήμα που ε, υπάρχει για τους σκοπούς αυτούς. Ακούσαμε τώρα τους τρεις ε, παρεμβαίνοντες, τον κύριο Στάικ, τον κύριο Χέλμπρεχτ και τον κύριο Βόλτερ. Ήρθε η στιγμή για ερωτήσεις και απαντήσεις. Προτείνω να ακολουθήσουμε την ε, συνηθισμένη διαδικασία. Για σκοπούς αποτελεσματικότητας λοιπόν, πρώτος γύρος ερωτήσεων, αφού πάρουν το λόγο ο εισηγητής μας, ο κύριος Κλοντ Μωράης και οι σκιώδεις εισηγητές, και μετά ένα πρώτο γύρο απαντήσεων από όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Οπότε μετά επιπλέον χρόνο για τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ και θέλουν να παρέμβουν ή να θέσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα ο συντονιστής μας, ο κύριος Κλοντ Μωράης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Ξέρετε, και εγώ Τώρα μόλις από λίγο αγόρασα μερικά αντιβιωτικά. Πάντως ε, άκουσα ότι είπε ο συνάδελφος από την Europol, διότι πρόκειται για ένα πάγιο θέμα το οποίο το έχουμε εδώ στις ακροάσεις μας όλοι, οπότε να μην σας εκπλήσει ε, το τι θα σας ρωτήσουμε όλοι εδώ. Γιατί ακριβώς γι' αυτό θέλουμε την Europol εδώ και το κέντρο κατά του εγκλήματος άκουσα αυτά τα οποία είπατε και πριν το τέλος της ομιλίας σας ε, είπατε ότι ε, τι έγινε με τους ισχυρισμού περί των υποκλοπών και είπατε ότι πρόκειται το κέντρο κατά του Ευρωεγκλήματος να αναλάβει την άμυνα κατά τέτοιων ε, υποκλοπών. Βέβαια το θέμα είναι ότι η Europol είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο και έχουμε ένα σωρό ισχυρισμού σχετικά με αυτά. Ας πούμε με την Belgacom, αποδείχθηκαν οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές. Ήρθαν εδώ πέρα ε, ανώτατοι πάλι να μας μιλήσουν. Δεν ήταν ισχυρισμοί, είναι αποδεδειγμένα γεγονότα περιστατικά. Απομένως, η ερώτηση μου είναι η εξής. Γιατί δεν κάνετε τις σχετικές ερευνές αν, θέλετε στο μέλλον να ε, μας προστατεύσετε ή να προστατευτείτε εσείς από υποκλοπές. Αυτό ήθελα και εγώ και άλλοι να να ρωτήσουμε. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο από την Ενίζα, αλλά και τον κύριο Βάλτερ. Τι γίνεται εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο για την πληροφορική μας. Ξέρω ότι ασχολείστε με κρυπτογράφηση και το σύστημά μας, αλλά για πες μας τι τι, τι γίνεται με το σύστημα του Κοινοβουλίου και την ασφάλειά του. Τι θα μας συνιστούσατε να κάνουμε. Επίσης μας μιλήσατε για αυτό το εμπορικό λογισμικό. Είναι ανοιχτής πηγής. Είναι καλύτερα σε αυτήν την περίπτωση. Τι γίνεται αν κανείς δεν έχει τέτοιες ε, λύσεις που είναι στο εμπόριο. Τι γίνεται όταν προέρχονται από τη είπα. Τώρα έχουμε με την ίδια σειρά τις απαντήσεις από τους προσκεκλημένους μας. Πρόεδρε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μωράης. ενώ κατά του κυβερνού εγκλήματος συγκροτήθηκε στα πλαίσια της Europol. Έχει συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένη εντολή, συγκεκριμένο στόχο. Βασικά, η δουλειά μας είναι να βοηθούμε τα κράτη-μέλη στις έρευνε τους κατά του σοβαρού ε, οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. και οι ερευνές μας οδηγούν σε ποινική δίωξη και ενδεχόμενη καταδίκη. Το θέμα δεν είναι βέβαια αυτό. Εκεί που εστιάζουμε κυρίως την προσοχή μας είναι τι γίνεται με το εργαμένο έγκλημα και πώς αυτοί οι εγκληματίες θα πάνε στην φυλακή. Αυτό είναι το έργο μας το οποίο πιστέψτε με προϋποθέτει μεγάλες προσπάθειες αντίστοιχο προπολογισμό. Από τότε που αρχίσαμε την ιστορική διαδρομή μας θα πρέπει να δείτε πόση πολλή δουλειά είχαμε και πόσο έχουμε πετύχει. Και τα κρατημέλη και εξωτερική μας εταιρεία κυρίως ε, Μα αναθέτουν ε, περιπτώσει κυβερνοεγκλήματο για το οργανωμένο έγκλημα σε σχέση με την, την παλαιότερη φάση στην οποία είχαμε περισσότερε ε, έρευνε που είχαν περισσότερο σχέση με εγκλήματα σε εθνικό επίπεδο. Κάποιε λίγε δεκάδε, α πούμε ε, συλλήψει, ενώ τώρα έχουμε εκατοντάδε. Άρα τώρα Έχουμε υποθέσεις πολύ πιο μεγάλες, έχουμε περιορισμένους ανθρώπινους πόρους και επομένως το θέμα δεν είναι σε ποιο πλαίσιο κινούμεθα και γίνονται αυτά. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες μας ορίζουν για τη δουλειά μας τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής ο κ. Κρίμα που δεν απάντησα εγώ αυτές τις ερωτήσεις ε, αλλάξτε, αλλάξτε. Απαντήστε στην άλλη ερώτηση. Να πω το εξή. Η Ενίζα δεν ε, ασχολείται με τα συστήματα πληροφορικής των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος τους ή άλλως για να το λύσω αυτό. Για το open source, για τα συστήματα open source. Το πρόβλημα θα μιλάμε για την ασφάλεια είναι πως η ασφάλεια είναι κάτι ε, το οποίο χρησιμοποιούν αυτοί οι οποίοι πουλάνε firewall, αντιβιωτικά κτλ. Και όχι για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αν είναι κανείς μια εταιρεία και πουλάει ένα προϊόν, το ερώτημα είναι γιατί εξοδεύεις λεφτά σε ασφάλεια πληροφορικής. Πώς εξοδεύεις σε ένα κινητό. Ε, πόσο σε ενδιαφέρει αν πουλάς αυτοκίνητα. Και δεν έχουμε βρει ένα μοντέλο ε, όπου είναι επιχειρηματικό μοντέλο εκεί όπου χρησιμοποιείται οριζόντια η ασφάλεια. Να σας πω, πριν από έξι χρόνια είχα μία συζήτηση με έναν άνθρωπο που ήταν επί δεκαετία ε, ε, υπεύθυνο για, την, για τα σύστηματα πληροφορική μια ασφαλιστική εταιρεία. Και τι έκανε αυτό ο άνθρωπο, IBM, Oracle, έτοιμα συστήματα κτλ. Στην ε, άλλη περίπτωση ε, που είχαμε μια υπηρεσία ασφαλείας συνέβη το εξής. Η μισή υπηρεσία δούλευε με Microsoft και η άλλη μισή με open source. Έτσι, και πονοκέφαλος μεγάλος. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς ακριβώς θα ενσωματώσουμε την ασφάλεια της πληροφορικής στο επιχειρηματικό μοντέλο γιατί είναι και παράγοντας κόστους. Κύριε Βάλτερ, θα συμφωνήσω με τον κύριο Χάλμπρεχτ πως η ασφάλεια είναι περισσότερο μια διαδικασία και όχι κάτι το οποίο θα αγοράσει κανείς και τελείωσε. Και συμφωνώ επίσης πως για αντιβιωτικά και για αυτούς που πουλάνε τέτοια πράγματα και φτιάχνουν φάργολ κτλ. Ε, για αυτούς είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Για τους υπόλοιπους είναι ένα κόστος και περισσότερο βάρος. Αλλά εσείς ως Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να αλλάξετε αυτή την ισορροπία γιατί να είναι βάρος και να κοστίζει περισσότερα για όλους. Τι κάνουν αυτές οι εταιρείε που πουλάνε λογισμικό. Λεφτά θέλουν να βγάλουν, θέλουν να πληρώνουν τους μετόχους τους, οπότε δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλεια. Γιατί η ασφάλεια κοστίζει λεφτά και κόπο. Οπότε αν θέλουν να πληρώνουν τους μετόχους τους, αγνοούν την ασφάλεια και σας δίνουν αυτό το οποίο εγώ λέω software της μπανάνας. Δηλαδή όταν σας το στέλνουν είναι μια χαρά καθαρό, αλλά δεν, είναι, δεν έχει οριμάσει και δεν είναι ασφαλές. Και υπάρχει ένας απλός οικονομικός λόγος γι' αυτό. Γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά και η ασφάλεια κοστίζει. Δεν βγάζει λεφτά σε μια εταιρεία. Εσείς όμως ως κοινοβούλιο μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Εάν βοηθήσετε... Κοιτάξτε, οι εταιρείε παραδείγματο χάρη λογισμικού δεν είναι αστικά υπεύθυνε ε, για το προϊόν του. Εάν σα πουλήσει ένας ένα αμάξι και δεν το έχει φτιάξει σωστά, είναι υπεύθυνη η ασφαλιστική εταιρεία. Πρέπει να κάνει ανάκληση, να το επισκευάσει μόνη τη κτλ. Αυτό κοστίζει. Άρα οι εταιρείε αυτοκινήτων κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε όταν φύγει το αμάξι από το εργοστάσιο να λειτουργούν τα φρένα γιατί αλλιώ έχουν ευθύνη. Εάν αγοράσετε software υπάρχει πάντα η αποποίηση ευθύνης που πρέπει να πατήσετε πριν ανοίξω πρόγραμμα που λέει το πρόγραμμα αυτό παρέχεται ως έχει χωρίς καμία ευθύνη του κατασκευαστή. Εάν αλλάξετε την αστική ευθύνη για το software η οικονομική εξίσωση πλέον για τις εταιρείε είναι διαφορετική. Έχουν αστική ευθύνη. Αν στέλνουν λοιπόν προϊόντα τα οποία δεν έχουν εξορισμού ασφάλεια και ιδιωτική ζωή, θα πληρώσουν παραπάνω μετά. Γιατί οι πελάτες θα το στέλνουν πίσω, θα πρέπει να το ξαναφτιάξουν κτλ. Και δεν μπορούν να δώσουν μετά μέρισμα στους μετόχους. Όσο δεν το κάνετε όμως αυτό, πάντα θα είναι το λογισμικό μπανάνα. Από εσά εξαρτάται. Μάλιστα, θα ακούσουμε ένα δεύτερο γύρο από τους και οσηγητές, η Σόφι Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους τρεις ε, κυρίους. Ομολογώ πως γέλαγα λίγο στην εισαγωγή της Europol όταν είπατε πως έχετε κουλτούρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων κτλ. Γιατί είναι δουλειά σας μετά σκεφτόμουν, μα αυτά λέει και η NSA. Αλλά δεν είχαν υπολογίσει τον ανθρώπινο παράγοντα, οπότε τώρα κάποιος θα ξέρασε όλα τα μυστικά. Έπαθα κατάθλιψη μετά από αυτά τα οποία λέει ο κύριος εδώ δίπλα μου. Γιατί φαίνεται πως ποτέ δεν υπάρχει αρκετή ασφαλή Γιατί ο προϋπολογισμός ε, και η εμπειρία που απαιτείται ε, είναι κάτι το οποίο έχουμε θέσει ξανά στην Επιτροπή μας. Αλλά νομίζω πως μία από τις δυσκολίες είναι η κοινή γνώμη, ειδικά αν δούμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ευχαρίστω να βγω και να πω πως χρειαζόμαστε περισσότερο προϋπολογισμό της Ένωσης. Οπωσδήποτε όμως είναι ένας σίγουρος τρόπος να μην ξανακλεγεί κανείς, έτσι. Πρέπει να πείσουμε για ε, ψηλότερο προϋπολογισμό και έχουμε και το γελίο σύστημα του επταετούς προϋπολογισμού αλλά τέλος πάντων πρέπει να το δούμε αυτό το οποίο είπατε. Αυτό το οποίο είπατε για την αστική ευθύνη με ενδιαφέρει. Γιατί κάνετε τη σύγκριση με τα αυτοκίνητα και τα φρένα των αυτοκινήτων. Αλλά εκεί πέρα ε, ε, μπορεί να ορίσει κανείς μια προδιαγραφή, είτε δουλεύουν είτε δεν δουλεύουν, έτσι. Ενώ και εσείς ο ίδιος είπατε πως οι απειλέ ασφαλές εξελίσσονται συνεχώς. Δηλαδή, αγοράζει κανείς ένα προϊόν το οποίο σε μια χρονική στιγμή ανταποκρίνεται, αλλά μετά, ε, ένα χρόνο μετά δεν θα το κάνει. Οπότε πράγματι μπορεί να θεωρηθεί η εταιρεία υπεύθυνη. Θα ήθελα να ακούσω το εάν ε, υπάρχουν όντως τέτοιες προδιαγραφές. Μετά, ένα άλλο που διάσα χτες στην εφημερίδα για την ε, υπόθεση Belgacom που μας απασχολεί, πως προσπαθούν να αφαιρέσουν το κακόβουλο αυτό λογισμικό και δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Εγώ είμαι άσχετη. Ένα τηλέφωνο έχω και ένα τάμπλετ, αλλά ε, δηλαδή μιλάμε για σοβαρά πράγματα, έτσι να προσπαθούν τόσο καιρό για να μην μπορούν να το σβήσουν. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, αν έχετε κάποια ιδέα του τι είδου συλλογισμικό μπορεί να είναι αυτό και ποιο μπορεί να είναι από πίσω και τέλο, Μια ερώτηση που δεν απευθύνεται σε κάποιον ιδιαίτερα, αλλά απορώ που συζητάμε την ασφάλεια των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν το ευαγέ αυτό ίδρυμα πριν από δύο εβδομάδες υπέστη hacking ε, από κάτι πάρα πολύ απλό από ό,τι κατάλαβα και η μόνη αντίδραση ήταν να κατεβάσουν την πρίζα. Έτσι, κατέβασαν την πρίζα του Wi-Fi και λένε να αλλάξετε το συνθηματικό σας. Ε, τώρα είμαστε ασφαλείς. Όχι, ακούγεται. Ναι, ναι, το υποψιαζόμουν, λέει η κυρία Ινετφέλντ, ότι αυτό θα λέγατε. Οπότε, ε, δηλαδή, άμα να συζητάμε για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορική, καλό είναι να έρθουν και οι δικοί μα οι υπεύθυνοι. Είχαν έρθει μία εβδομάδα πριν μάθουμε για την προσβολή του συστήματό μα και μα λέγανε όλα μια χαρά. Και μάλλον δεν ήταν όλα μια χαρά, ίσως πρέπει να τους ξαναφέρουμε εδώ. Μάλιστα, ας ακούσουμε τώρα τους προσκεκλημένους μας. Απαντήσεις. Ότι γνωρίζω. Είχε συμμετική σχέση ο κύριος Σνόντεν. Τον είχαν αναθέσει κάτι με σύμβαση. Σας το είπα αυτό στην εισήγησή μου. Όμως ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν έχουν πρόσβαση στο λειτουργικό, ούτε στα, στα, στα, στα δεδομένα μας αυτά τα εσωτερικά. Είναι ξεκάθαρα οριοθετημένο τι μπορούμε να κάνουν και συμφωνώ. Όπως το είπατε. Όπως είπε εδώ και ένας άλλος προσκεκλημένος. Δεν υπάρχει 100% ασφάλεια. Απλώ θα πρέπει κανεί να έχει επίγνωση του τι γίνεται και να θωρακιστεί μέσα σε λογικά όρια όσο μπορεί περισσότερο. Και πάλι μπορεί κάτι να πάει στραβά. Δεν το αποκλείω για κανένα οργανισμό ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό σας τονίζω. Πάντω εμεί ε, όντω έχουμε αυτό το πνεύμα, αυτή την κουλτούρα τη ασφαλεία. Και οι συναδελφοί διορθώνουμε στον άλλο όταν κάποιος ε, κάτι παραλείψει όσον αφορά τα καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια. Οπότε γι' αυτό σας λέω θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα υψηλά όσον αφορά την ασφάλεια. Και επίσης... Ναι, ναι, καλά τα είπατε και για τα φρένα αυτοκινήτων και αν δεν λειτουργούν τα φρένα στο αυτοκίνητο δεν θα πρέπει κανείς να το χρησιμοποιεί. Το ίδιο ισχύει ότι αν υπάρχει κάποιος ε, ιός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο υπολογιστής, όμως γίνεται το αντίθετο. Ακόμα και όταν μου λένε ότι υπάρχει ιός, συνεχίζω και τον ε, χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου χωρίς να φέρω ευθύνη εναντί των άλλων συναδέλφων. Μα γιατί θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά την ασφάλεια των υπολείπων, των συναδέλφων. Θα έπρεπε κάποιο να πει άπαρχη έχει ιό κάποιο υπολογιστή, τέρμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και να, ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να μα απασχολήσουν. Η ευθύνη όχι μόνο του κατασκευαστή αλλά και του χρήστη. Um, a general statement. Uh, κάνω μια γενική παρατήρηση. Εδώ έχω αυτό το smartphone, λέει ότι έχει το σύστημα Android. Δηλαδή, το κλείνω τελείω. Άρα το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο αναφέρατε όσον αφορά την πρικοδότηση. Λέει ο κύριος Το πρόβλημα είναι η τεχνολογία μας ε, είναι τέτοια, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι και Κοιτάξτε, το διαδικτύο ξεκίνησε με πάρα πολύ απλά πρωτόκολλα και πρότυπα. Όμως, τις 20-30 χρόνια ε, αρχίσαμε να ασχολούμεθα με την ασφάλεια και το πρόβλημα είναι ότι όλοι χρησιμοποιούν όσο γίνεται περισσότερη ασφάλεια και κρυπτογράφηση κλπ. Όπως μου είπε τώρα λοιπόν το smartphone κρατάω. Ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να φάει έναν ιό, να είναι να του υποκλέψουν τα δεδομένα, ε, τα password κλπ. Οπότε ναι, μπορεί να αλλάξει το password, αλλά το πρόβλημα είναι πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Ναι, δεν οδηγούμε γρήγορα όταν είναι ολισίρο το δόστρωμα, αλλά το κάνουμε με τα gadget, με τους, με Άρα είναι το θέμα επομένω της διακυβέρνησης, της χρήσης των gadget. Ε, τέτοιο παιδί χρειάζεται και οπότε το θέμα είναι να εκπαιδεύσουμε τους ε, χρήστες για να ξέρουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Um, first... Πρώτα απ' όλα, για την πρώτη ερώτηση που δεν απάντησα, για το software open source. Μπορεί τουλάχιστον κανείς να δει τι κάνει ακριβώ το software, γιατί έχει τον κωδικό. Και σε περίπτωση κατεπήγοντο μπορούν να τα φτιάξουν οι υπηρεσίε σα γιατί έχουν τον κωδικό. Ενώ στα εμπορικά συστήματα υπάρχει ένα μαύρο κουτί του οποίου δεν έχετε ιδέα και γνώση το τι κάνει. Όταν είχα ξανάρθει στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν δύο εβδομάδε, τα έχετε πει και προηγουμένω. Ανθρώπινο παράγοντα, αυτό είναι το πιο απρόβλεπτο στοιχείο. Αλλά και οι τεχνικοί παράγοντες. Εάν κατάλαβα καλά την επίθεση που έγινε, υπάρχει ε, ένα ασύρματο σύστημα για προσκεκλημένους και κάποια μέλη το χρησιμοποιούσαν ε, για να συνδεθούν στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, στο email τους. Κάποιοι λοιπόν μπόρεσαν να πάρουν τα, τους κωδικούς και τους, τα ονόματα χρήστη για να συνδεθούν στο mail τους. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα, το δημόσιο, στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε να ε, συνδεθεί και να πάρει τα δεδομένα για να μπουν στο mail τους. Αυτός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και το άλλο είναι ότι το τμήμα IT σας δεν φρόντισε. Δεν φρόντισε οι πελάτες ε, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, των, της ταμπλέτας, οτιδήποτε, να έχει πρώτα ένα κωδικοποιημένο διάβλο. Αν έχετε WPM, στην έναρξη αυτομάτως δεν γίνεται γιατί μπορεί κανείς να πάρει στοιχεία από την κίνηση ενός λογαριασμού αλλά όχι το όνομα χρήστη και τον κωδικό γιατί είναι κωδικοποιημένα όλα αυτά. Εάν έχει γίνει σωστά η κωδικοποίηση και δεν μπορεί κανείς να πάρει τα αρχικά στοιχεία για την κωδικοποίηση, τουλάχιστον αυτό δεν παραβιάζεται από ένα 14χρονο. Ή τέλος πάντων όποιον ε, και αν σκεφτούμε ότι μπορεί να ήταν. Αυτό που είπε προηγουμένως είναι ότι οι επιτιθέμενοι συνήθως ξέρουν το δίκτυο στο οποίο παρισφρίουν πολύ καλύτερα από τους ε, αμυνόμενους. Εάν κάποιος έχει 100 ή 1000 συστήματα ως ένας administrator, ο hacker διαθέτει πολλά πρόσωπα με ιδιαίτερες δεξιότητες για να επιτεθεί σε ένα και μόνο σύστημα και όλοι συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους για αυτόν τον σκοπό. Συχνά υπάρχουν φήμες ότι οι hackers φτιάχνουν έτσι το σύστημα στο οποίο παραβιάζουν, ώστε να μην μπορέσουν οι διαχειριστέ του σύστηματος να το κοιτάξουν πολύ προσεκτικά. Ω hacker λοιπόν κανεί αυτό μπορεί να κάνει καλά είναι να αφήσει το σύστημα να λειτουργεί. Διότι δεν το παίρνουν χαμπάρι οι διαχειριστέ και δεν προσέχουν τι συμβαίνει δεν ε, μου κάνει εντύπωση που δεν μπορείτε να απομακρύνετε αυτό το malware, γιατί έχουν καλύτερα, περισσότερα λεφτά οι hackers, έχουν περισσότερε δεξιότητε και ικανότητε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, έναν δυνάμει του περισσότεροι, ενώ εσεί από την άλλη έχετε έναν administrator, έναν διαχειριστή, ο οποίο πρέπει να φροντίσει δεκάδε, εκατοντάδε ή χιλιάδε συστήματα ταυτόχρονα. Πόσο στενά μπορεί να παρακολουθεί το κάθε σύστημα, πόσο στενά, ε, πόσο καλά μπορεί να ξέρει το σύστημα, πόσο καλά καταλαβαίνει τεχνικός τι συμβαίνει στο σύστημα. Και ίσως και το εμπορικό ε, σύστημα που χρησιμοποιεί το λογισμικό να έχει ένα μαύρο κουτί. Ένα μαύρο κουτί που το έχει φτιάξει ο κατασκευαστής. Δεν σημαίνει ότι μπορεί ο διαχειριστής να κάνει όσα το σύστημα υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρετε τι δίωδη, ε, τι κερκόπορτες υπάρχουν από τις εταιρείες που κατασκεύασαν το σύστημα εκτός Ευρώπης. μπορεί να υπάρχουν παραβιάσεις ή επιδράσεις από αντιπάλους στην κατασκευή. Ακόμη λοιπόν και αν αλλάξετε το λογισμικό μπορούν να μπουν ξανά την επόμενη μέρα διότι έχουν ένα μυστικό κωδικό που μπορεί πάντοτε να τους ε, αναγνωρίζει. Ίσως από το εργοστάσιο να είναι φτιαγμένη αυτή η κερκόπορτα. Αν έχετε λογισμικό open source τουλάχιστον μπορείτε να τη βρείτε αυτή την κερκόπορτα. Και συνήθως δεν είναι καν ε, μια κερκόπορτα, είναι ένας... Ε, είναι ένα μικρό σύστημα, μια, ένα σφαλματάκι, έτσι παρουσιάζεται αυτό το σύστημα, ένα bug όπως λέγεται, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για κερκόπορτα. Όταν λοιπόν δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει τις πραγματικές κερκόπορτες, εντοπίζει αυτά τα bugs και το σύστημα αποτυγχάνει. Αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε στους επόμενους, τους σκιώδες εισηγητές. Κύριε Άλμπρεχτ, έχετε το λόγο για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω πρέπει να γίνω λίγο πιο επιθετικός με τους προσκεκλημένους μας, ξεκινώντας με τη Europol. Διότι εσείς ε, μας είπατε ότι πρέπει να επικεντρωθείτε και να το καταλάβουμε κι εμείς ότι επικεντρώνεστε στο οργανωμένο έγκλημα και τα όσα περιλαμβάνει η εντολή σας. Εάν κοιτάξω την ετήσια έκθεση της Europol, τι βλέπω. Τρομοκρατία. Σας ε, απασχολούν αυτά κυρίως. Τόσα θέματα στις εκθέσεις σας. Ε, και εδώ μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις Για να μην πω για κυβερνοπόλεμο. Κυβερνοπόλεμο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από επιτιθέμενους που δεν τους γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε ποιος τα υποκίνησε όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν να αποκλειστεί ότι πρόκειται για εγκληματία ή για μια αρχή που δρά εκτό νόμου δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί αν δεν υπάρξει έρευνα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όμω πρόκειται για επίθεση και δεν είναι μια μικρούλα επίθεση. Είναι ε, μια επίθεση όπως αυτή κατά της Μπέλγακομ. Ήταν τεράστιο αυτό. Ε, επίθεση που αποδείχθηκε από τον Σνόντεν με έγγραφα κατά μια υπηρεσίας ε, και τη Yahoo και τη Google. Έχουν αποκαλυφθεί σήμερα με δεδομένα οι κινητές επικοινωνίες με συγκεκριμένες ε, ταυτότητες έχουν ε, αποκαλυφθεί, ήταν ε, προσβα, προσβάσιμες καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τεράστιο όγκο και εδώ μιλάμε αδίκημα και παραβίαση του ποινικού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων ψηφίσαμε πέρσι για το κυβερνοέγκλημα. Και θα πάω και παραπέρα. Ο Σνόντεν Μα έδωσε και οικονομικά πολύτιμε πληροφορίε, για παράδειγμα. Τι υποκρύπτουν όλα αυτά, την τεράστια τιμή όλη αυτή τη υπόθεση. Μιλάμε για δισευρώ. ευρώ. Εδώ <clears throat> δεν μιλάμε απλώ για οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για οικονομικό έγκλημα που πρέπει να καταπολεμηθεί. Έγκλημα κατά της ασφάλειας των πληροφοριών. Και των δικαιωμάτων των πολιτών βεβαίως, αλλά αυτό δεν είναι καν τόσο σημαντικό έτσι όπως τα βλέπετε εσείς τα πράγματα, προφανώς. Όταν λοιπόν τα συζητάμε αυτά, πραγματικά νομίζω ότι θα έπρεπε να διορθώσετε τις προτεραιότητές σας. Εγώ είχα την εντύπωση ότι δαπανίσαμε χρήμα για το EC3. Ναι, Βεβαίω προβλέψαμε επιπλέον κονδύλια από τον προπολογισμό μα για τη Europol. Μάλιστα, ε, διατέθηκαν κονδύλια για το EC3. Και ήμουν υπέρ και ακόμα είμαι υπέρ. Αλλά σας παρακαλώ, τουλάχιστον κάντε σωστά τη δουλειά σας. Εδώ μιλάμε για ε, εγκλήματα, αδικήματα που έχουν να κάνουν με κυβερνοϋποθέσεις. Ερευνήστε τις κυβερνοϋποθέσεις, ε, επιθέσεις. Υπήρξε οποιαδήποτε αρχή, οποιοδήποτε ε, τους μέλους που να ζήτησε τη βοήθειά σας για να ερευνήσετε πιθανές παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης, πιθανές παραμβιάσεις όπως τις ορίζει ο ποινικό μας κώδικας ή οι νομη μας. Εάν όχι, και πάλι είναι απαράδεκτο σε σχέση με τα περιστατικά της Belgacom. και την πρόσβαση σε εταιρείε τηλεπικοινωνίας άλλων κρατών μελών, αλλά και το τι γίνεται με εκατομμύρια, με τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών, ε, εκατοντάδες εκατομμύρια πολιτών. Αλλά το θέμα δεν είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα μόνο και κυβερνά ασφάλεια, αλλά και το θεμελιώδες δικαίωμα της, ε, του απορρίτου και της ε, ε, μυστικότητας των επικοινωνιών μου. Μιλάμε για θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη. Πραγματικά λοιπόν αναρωτιέμαι εάν το καταλαβαίνετε αυτό στα κεντρικά σας και πραγματικά θα ήθελα ενεργά να κάνετε κάτι, να προωθήσετε αυτές τις έρευνες. Ρωτήστε τις αρχές των κατομελών Δεν πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες. Όταν μιλάμε για το SWIFT, όταν μιλάμε για την ε, ευρεία πρόσβαση στα δεδομένα SWIFT παρά το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε έρευνες από αυτού. Και αν δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα, μιλήστε εσείς με τι αρχέ. Μιλάμε για καταπολέμηση εγκλήματο. Πραγματικά, τι κάνουμε εδώ πέρα. Αυτά για την Europol και με συγχωρείτε που χασούμερισα τόσο <clears throat> για την Ενίζα. Και εδώ πρέπει κάτι να διορθώσουμε στην ε, οπτική μας γωνιά. Για ποιο σκοπό ε, δημιουργήσαμε την Ενίζα. Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εδώ καλύπτουμε ε, και την προστασία κάθε πληροφορίας και συστήματος πληροφοριών στην Ευρώπη και ελπίζω και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως αν μιλάμε για το CRT. Με τις ομάδες που θα έπρεπε να αντιδράσουν στις επιθέσεις και το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να είναι στο κέντρο της προσοχής σας. Αλλά αν δεν θέλετε να μιλήσετε για αυτά, ας μιλήσουμε για τα συστήματα της Microsoft. Σε όλα τα δίκτυα των θεσμικών μας οργάνων. Προφανώς υπάρχουν τεράστια παραθυράκια. Οποιοςδήποτε hacker μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό μου email, στο λογαριασμό μου, μέσα του συστήματος της Microsoft και να πάρει το περιεχόμενο των email. Ε, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Για επικεντρωθείτε λίγο σε αυτό. Εσείς πώς το βλέπετε. Πώς βλέπετε αυτά τα παραθυράκια, πώς μπορούν να καλυφθούν. Και τι χρειάζεται από την πλευρά των πολιτικών, των πολιτικών συνόντων να αλλάξει. Εάν θεωρείτε ότι θέλουμε να πετύχουμε την πραγματική ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και τελευταία μου ερώτηση προς τον κύριο Βάλτερ. Για τα παραθυράκια από το ότι υπάρχουν, τι κλικόπορτε. Ε, εσείς γνωρίζετε στην Πέλγα ακόμη, σε άλλα συστήματα επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και των σχετικών του πληροφοριών. Γνωρίζετε τι δίκτυα χρησιμοποιεί η Ευρώπη. Ξέρετε συγκεκριμένε κλικόπορτες, τι γνωρίζετε. Διότι υπονοήσατε ότι υπάρχουν αυτές. Υπάρχει κάποιος που ασχολείται με αυτές, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Με τη δουλειά της ενίσα ενδεχομένως. Μπορείτε να μας δώσετε μια εσωτερική εικόνα του τι συμβαίνει με αυτά. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε έτσι στην Επιτροπή Ελευθεριών, οπότε οπωσδήποτε μπορεί ο καθένας ελεύθερα να πει την άποψή του για το κάθε θέμα, αλλά επειδή έχουμε τρία θέματα το απόγευμα αυτό και περιορισμένο χρόνο, σας παρακαλώ να μείνετε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε κάποτε γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, ο, τώρα είναι η ώρα των απαντήσεων. Κύριε Μπύρχερ Κοιτάξτε. Έχετε, έχετε δίκιο. Εμεί πάντα με ανοιχτό μυαλό κοιτάμε τις υποθέσεις. Έχουμε διάφορες υποθέσεις. Ε, τεράστιες υποθέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και βοηθάμε τα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν καλύτερα τους πόρους τους. Συνεισφέρουμε με εργαλεία, Τώρα πλέον έχουμε και εξουσίες, ε, μπορούμε να πάμε στα δικαστήρια, ε, στο, στο, στα εθνικά και στο ΔΕΚ και στα εθνικά δικαστήρια, εθνικές εισαγγελίες κτλ. που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία. Έχουμε επίσης την δυνατότητα να ζητήσουμε από κράτη-μέλη να εξετάσουν κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν δούμε πως κάποια πράγματα ε, γίνονται από κράτη Εάν είναι οργανωμένο το έγκλημα βεβαίως το κυνηγάμε, αλλά όταν ε, κάτι είναι ε, από κράτη υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν. Πρώτα απ' όλα, ε, γι' αυτό έχει συσταθεί η ομάδα μας. Μα μιλήσατε για κυβερνοπόλεμο. Ο κυβερνοπόλεμος είναι αρμοδιότητα του στρατού μετά, έτσι. Είναι αλλού δουλειά. Μετά, κρατικές επιθέσεις κατά κρατών. Ε, μετά μιλάμε για εθνικό επίπεδο. Ε, αυτό αφορά τις εθνικές υπηρεσίες μετά, όχι τις αστυνομίες. Οπότε εμείς ασχολούμαστε κυρίως με αστυνομίες ε, και ο στόχος είναι να έχουμε κάτι το οποίο θα σταθεί σε δικαστήριο για να επιτύχουμε καταδίκη. Και επειδή, ε, λόγω των πραγμάτων που βρήκαμε, επειδή ο κύριος Σνόντεν ε, είπε κάποια πράγματα, εξορισμού υποθέτουμε πως είναι κάτι με στήριξη κάποιου κράτους. Οπότε, πού εστιάζουμε εμείς. Αυτό το οποίο κάνουμε κατά βάση είναι να δούμε ε, το, αυτό το οποίο μας λένε τα κράτη-μέλη. Έχουν τα κράτη-μέλη τις εξουσίες για να ερευνήσουν και αυτές παίρνουν τις αποφάσεις τι θα ερευνηθεί και τι όχι έτσι και τέλος αποφασίζουν το εάν θα εμπλέξουν την ε, Europol και το δικό μας το τμήμα. Οπότε γι' αυτό με βάση αυτά τα οποία είδαμε ε, μας ζητάνε τα κράτη-μέλη να τα βοηθήσουμε και να δούμε την ε, ζημιά που γίνεται και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Εάν δείτε τη ζημιά που γίνεται γενικά από το κυβερνοέγκλημα στην οικονομία, εμείς υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη ένεργα, αλλά όταν μιλάμε για πράγματα τα οποία τα στηρίζουν κράτη-μέλη, δεν, έχουν, ε, δεν θέλουν τα κράτη-μέλη η εμπλοκή της Europol. Ε, τότε πρέπει να σα ρωτήσω δύο πράγματα συγκεκριμένα. Πρώτον, σημαίνει αυτό πως ξέρετε, αποδείξατε δηλαδή πως αυτές οι επιθέσεις ήταν με στήριξη κράτους. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η Europol ε, δεν το ψάχνει. Γιατί ξέρετε πως είναι με την υποστήριξη κράτους. Και δεύτερον, Είχατε αιτήματα από κράτη-μέλη να ερευνήσετε τις επιθέσεις αυτές ε, σε στήματα όπως της Belgacom, Swift, Yahoo κτλ. Για το ε, πρώτη ερώτηση, ακόμα δεν έχουμε δει υποθέσεις ε, τέτοιες, δηλαδή να ξεκινήσαμε εμείς από το μηδέν και να διαπιστώσαμε ότι είναι κράτος μπλεγμένο και να το αναπέμψαμε, δηλαδή θα το ήξερα, για τη δεύτερη ερώτηση δεν είμαι απολύτως σίγουρος, δεν ξέρω το εάν ε, ε επισήμως ή ατύπως μας έχει δίσει κάποιος βοήθεια για την Belgacom τη SWIFT. Δεν μου λέει τίποτα και εγώ είμαι υπεύθυνο ε, της στρατηγικής, ε, αλλά άλλος είναι υπεύθυνο για το κομμάτι επιχειρήσεων. Αλλά, μάλλον να το πω αλλιώς, θα, κάτι θα ήξερα, είναι πιθανό να το ήξερα αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ να σα το πω 100% αυτή τη στιγμή. Και τώρα, καθηγητά, έχετε εσεί το λόγο. Ναι, ναι, καταλαβαίνω 100% το οποίο να πείτε όμω για μα η πρόκληση ω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είναι το εξή, ότι έχουμε μια καινούργια εντολή φέτο και ε, σε αυτή τη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο ε, δεν ήθελαν να μας δώσουν κάποιο είδους καθήκοντα επιχειρησιακά έτσι απλά. Και επίσης έχουμε τον κονισμό μας που θα αξιολογηθεί πάμε στο 18 για το Κοινοβούλιο είπαμε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε συστάσεις. Και όσον αφορά το θέμα της συζήτησής μας για την παρακολούθηση και τις υποκλοπές, τα κράτη-μέλη προσέχουν τόσο ώστε αυτά τα οποία μας απασχολούν να μην έχουν να κάνουν καθόλου ή τελικά να μην ε, αγγίζουν, μην, μην θίγουν την εθνική κυριαρχία. Για αυτά τα κενά, τα παραθυράκια στην ασφάλεια, τις κερκόπρωτες, όπως είπαμε, φυσικά ε, δεν είναι αυτό ο σκοπός, ούτε κανένας το δηλώνει ότι έχετε τέτοιο είδους γεργόπορτα και ουδέποτε επομένως εκουσίως υπάρχουν τέτοια, τέτοια χαρακτηριστικά εγγενή στο σύστημα, ούτω ώστε να λειτουργήσουμε τον τρόπο που είπατε. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο περιπτώσεις και τις οποίες τις γνωρίζουμε από, το, από την υπόθεση Έσσελον πριν από μια δεκαετία και θυμάμαι ότι το API κάποιος αυτό τον κώδικα κλειστής πηγής, τον ανέλησε, τον έσπασε. Και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουν ε, μια άλλη εκδοχή με τα σύμβολα, τα αντιβιωτικά. Είχαν βάλει ακόμα και τίτλους. Μπορούσε κανείς να δει τι περί τίνος και τελικά αυτό το οποίο βρέθηκε τότε στα, σε αυτήν την εκδοχή των Windows ήταν ότι υπήρχε και ένα δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης το οποίο λεγόταν NSA.key έτσι λεγόταν. άρα αυτό τι έκανε αργότερα η Microsoft ότι αυτό ήταν για backup, αλλά βέβαια αυτά όλα είναι βλακίες. Δεν χρειαζόταν εκεί πέρα να υπάρχει τέτοιου είδου ε, ε, κλειδί ε, για backup. Θα μπορούσε να υπάρχει, να υπάρχει το ίδιο κλειδί σε δύο διαφορετικά μέλη. Οπότε, για να ρωτήσετε και εσείς μόνοι σας, γιατί να υπάρχει ένα τέτοιο κλειδί και να λέγεται NSA.key. Το συμπέρασμα δεν μπορεί παρά να είναι το προφανές. Αλλά σας αφήνω το σκεφτείτε για μόνοι σας. Τώρα ένα άλλο παράδειγμα μπορώ να σας δώσω. Είναι ένα πρόγραμμα της IBM. Είχαν κάτι το οποίο το, το λέγανε ακόμα και στα, στους, στους οδηγούς χρήσης, τους Και είχε να κάνει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Και είχε εκεί πέρα τα κομμάτια του, του, του, της, του, της αποκρυπτογράφησης τέλος πάντων εκεί πέρα και αυτό ήταν κρυπτογραφημένο με, με κάποιο άλλο είδους ε, κλίδα. Οπότε με αυτή την κλίδα θα μπορούσε κανείς να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα email και λόγω αυτού του χαρακτηριστικού μπορούσε κανείς να τα, να τα αποκρυπτογραφήσει. Άρα μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει το κάθε mail, το κάθε μήνυμα. Οπότε και εδώ μπορούμε να βρούμε τι ωφελούσε αυτή η κλίδα. Αν αυτό το έδινε κανεί σε υπηρεσία πληροφοριών, σε διοικητική αρχή, τότε θα μπορούσαν εκείνοι να διαβάσουν όλα τα κρυπτογραφημένα email του συστήματο, ενώ, ενώ οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να τα διαβάσουν. Άρα, βλέπετε εδώ πέρα κάποιε ενδείξει σαφέ σε σχέση με το πώ ε, εφαρμόζονται, πώ υλοποιούνται, πώ χρησιμοποιούνται αυτές οι κερκόπορτες. Οπότε οι αντίπαλοι μας βέβαια ε, και, και αυτοί αντλήσαν συμπεράσματα, οπότε δεν κάνουν τόσο φανερά πράγματα. Τα ρούτερ ας πούμε. Αυτά τα οποία στέλνουν ε, με τα κινητά, με το ίντερνετ, τα, τα δεδομένα μας. Αυτά τα κουτάκια που τα λένε router, routers. Στα ε, και, για κοιτάξτε τι γίνεται με την ασφάλεια, με το Google. Έχουν τόσο, τόσα, τόσα, πολλά μολυσματικά στοιχεία, τόσο αυτός πολυσιούς εκεί μέσα. Πάρα πολύ εύκολο. Με ε, κάποιον έτσι εκπαιδευμένο λίγο και λίγα λεφτά, κανείς μπορεί να τους το αναθέσει και να τα διαλύσουν αυτά τα ρότερα. Ακόμα και hacker που δεν έχουν λεφτά θα μπορούσαν εκεί σε λίγες εβδομάδες να βρουν τρόπους ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν ό,τι θέλουν και να, να, να, να ε, υποκλέψουν τελείως αυτό το λέει. αυτό το πει σε κάποια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών. Ότι ότι, ότι, ότι, ότι μπορεί να ελέγξει χιλιάδες ρούτερ μέσα σε ένα δίκτυο, τότε τι. Δεν μπορεί κανένας να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι κακό θέλει με αυτό. Έχουμε ξεφύγει πολύ από το πρόγραμμα, αλλά ακόμη ζητούν το λόγο οι σκιώδεις. Ε, σας παρακαλώ, κοιτάζετε την ώρα, γιατί έχουμε ακόμη δύο πάνελ. Πρόεδρε, Κυρία Ένστ, ναι, κύριε Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όντως δίνει περισσότερα λεφτά για χαρτί υγείας από ό,τι για την ασφάλεια της πληροφορικής. Έτσι. Έχω καταλάβει σωστά ή όχι. Έχουμε υποτίθεται πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που εγκρίναμε, στο οποίο ε, κάναμε περικοπές από εδώ και από εκεί ε, έτσι, με πολύ ορμή. Οπότε, τι έχουμε τώρα, 7 χρόνια μπροστά μας ε, μέχρι το 2020. Ε, καλό να μην ελπίζουμε σε ασφάλεια της πληροφορικής γιατί δεν υπάρχουν λεφτά και περικόπηκαν κιόλας. Οπότε όλα αυτά τα οποία λέμε είναι θεωρίες, ωραίες θεωρίες αλλά χωρίς αντίκρισμα. χρειαζόμαστε πράγματι ικανούς συνεργάτες που θα αντιλαμβάνονται τις αλλαγές και βεβαίως με πράγματι ένα άτομο δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά αλλά Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί στις ε, είπα Είχα λάβει κάποια σχετικά email, ε, παραδείγματο χάρη ε, και μετά βλέπουμε ε, το συμβάν που έγινε εδώ πέρα που μου λένε κάποιον συνάδελφο υποκλέψανε και αλλάξτε το συνθηματικό σας. Ε, πρακτικά, τι θα κάνω εγώ ως βουλευτής, πώς θα προστατευτώ. Δεδομένων των πραγμάτων, έτσι, που έχουν όπως έχουν. Και μου είπατε πως ε, αν δεν ξοδέψουμε πολλά εκατομμύρια δεν πρέπει να έχουμε και καμία ελπίδα για να αντισταθούμε. Δεύτερον, Europol. Κατάλαβα σωστά, όντως δεν ξέρετε αν έχουν υπάρξει περιστατικά συμβάντα ή όχι. Αυτό είπατε, ότι δεν ξέρετε όντως αν έχει γίνει κάτι. Ήρθε η ώρα για απαντήσεις, ε, κύριε Μπίρχερντάικ. Κατάλαβα καλά. Κυρία Ένστ, μιλήσατε για την προηγούμενη απάντησή μου που είπα ότι δεν ε, ξέρουμε... Ναι. Το πρόβλημα είναι πως ε, εάν δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς συζητάει δεν μπορεί να καταλάβει αν τον έχουν χακάρει. Έτσι. Υπάρχουν κάποια εμπόδια ε, μετά, εάν ε, υπάρχει κάποια παράξενη συμπεριφορά μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς μπορεί να φροντίσει το προσωπικό του να αξιολογεί τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα μέτρα που μπορούν να ληφθούν αλλά 100% σιγουριά και εγγύηση δεν υπάρχει ότι είναι κανείς δηλαδή απολύτως ασφαλής. Οπότε, δεν υπάρχει 100% εγγύηση. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να προλάβουμε κάτι και να ανοιχνεύσουμε αν έχει συμβεί. Ε, ό,τι μπορεί να γίνει το έχουμε κάνει, αλλά αυτό ισχύει για όλους, έτσι. Γιατί δεν κοιτάω κάθε μέρα κάτω από το αυτοκίνητό μου να δω πως μου έχουν βάλει συσκευή παρακολούθησης, γιατί δεν, τι να πω, δεν το περιμένω έτσι. Αλλά εάν γνωρίζει κανείς πως υπάρχει αυτή η απειλή θα το έκανε κάθε μέρα. Και αν το βάζει κάθε μέρα σε κλειδωμένο γκαράζ το αμάξι, ήδη ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Απαντήσω γερμανιστή. Βεβαίω. Ε, κοιτάξτε, α είμαστε λίγο ήρεμοι έτσι. Ψυχραιμία. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κάνουν πάρα πολλά ε, για την ασφάλεια και δίνουν, μην ανησυχείτε, δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά για την ασφάλεια της πληροφορικής από ό,τι για το χαρτί του αλέτας, τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε. Α, ρωτάτε τώρα το τι μπορείτε να κάνετε. Υπάρχει μία σύσταση της ΕΝΙΖΑ που μπορείτε να εφαρμόσετε για τα κοινωνικά δίκτυα, τι κάνουμε με τις ε, μικροεφαρμογές της <laughs> τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να υπογράψω το ε, email μου και να το κωδικοποιήσω, το PGP για τον απλό χρήστη, για την κωδικοποίηση εγώ θεωρώ πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο αυτά τα οποία έχουμε και αυτό γιατί ε, αυτά που έχουμε δεν τα χρησιμοποιούμε ήδη αρκετά ας χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε και μετά μάλιστα κύριος βάλτε; μια που εγώ δεν ξέρω την ε, τεχνολογία που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν ξέρω πώς αξοδεύεται για χαρτί υγείας και ασφαλεία. Σε μεγάλους οργανισμούς πάντως περισσότερα πάνε στις τουαλέτες. Εν πάση περιπτώσει. Ίσως οι πόροι διαθέσιμοι για την πληροφορική και την ασφάλεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά για να δείτε τα ζητήματα τα προφανή. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε κανονισμούς που έχετε σε περισσότερους, περισσότερους μεγάλους οργανισμούς οι χρήστες, εσείς είστε χρήστες δεν μπορούν να εγκαταστήσουν PGP στον υπολογιστή γιατί δεν έχετε ε, προνόμια διαχειριστή δεν σας ανήκει τελείως ο υπολογιστής σας, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εσείς ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε σε ένα διαχειριστή και να πείτε θέμε να βάλουμε PGP και κάντε μας για μια εκπαίδευση ή να πάρετε την άδεια να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Κάτι άλλο. Είναι βεβαίως να εκπαιδεύσετε τους χρήστες. Τον ανθρώπινο παράγοντα. για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για τα ασύρματα δίκτυα, wireless LAN κτλ. Εδώ πέρα δηλαδή ήταν σαφές ότι ήταν ο ανθρώπινος παράγοντος. Κάποιος έστειλε τα διαπιστευτήριά του, τα συνθηματικά και το όνομα χρήστη, χωρίς κρυπτογράφηση σε ανοιχτό δίκτυο, έτσι. Αν τώρα μάθατε λοιπόν πως αυτό είναι επικίνδυνο και μπορεί ο καθένας να δει τα συνθηματικά σου, δεν το κάνουμε από εδώ και μπρο. Το πρόβλημα είναι πως ο κόσμος δεν έχει ιδέα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα και το τι κάνουν ε, ανά πάσα στιγμή, έτσι. Οπότε, ε, τι να πω, εκπαιδεύστε καλύτερα τους χρήστες. Φροντίστε να τους ε, κάνετε να καταλάβουν τι κινδύνους αντιμετωπίζουν, έτσι. Ακούσαμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις και κανονικά θα πρέπει να έχετε την ε, δυνατότητα να κάνετε και άλλες ερωτήσεις, αλλά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στον χρόνο, οπότε πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή στο επόμενο θέμα, το οποίο αφορά την παρουσίαση από τον κύριο Μωραέ στο εγγράφο εργασίας για την παρακολούθηση από αμερικανικές υπηρεσίες και ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Και θα μας πει τι έγινε με την αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Μωραές. Κύριε Μωραές, έχετε το λόγο. Και βεβαίως, αποχαιρετάμε τους καλεσμένους του πρώτου πάνελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο μας είπατε. Ευχαριστώ. Thank you, thank you, thank you. Now, Mr. Moraes, floor yours. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι έχουμε φύγει πολύ εκτός προγράμματος. Συνάδελφοι προσκεκλημένοι, ξέρω ότι όλοι έχετε τρένα να προλάβετε πτήσεις. Θα είμαι λοιπόν τάχιστος. αλλά δεν έχω την πρόθεση να μειώσω τη σημασία οποιοδήποτε θέματος. Απλώς πρέπει να βιαστούμε. Διότι έχουμε πέντε έγγραφα εργασία που πρέπει να καλύψουμε. Θα ήθελα σε αυτό το τμήμα της συζήτηση, Πρόεδρε, να μιλήσω για το έγγραφο εργασία, για την παρακολούθηση και μετά αυτό που είχαμε στην Washington και μετά να έχουμε ερωτήσεις. Οργανώστε το όπω θέλετε. Ωραία πάμε στο έγγραφο εργασία για τι πρακτικέ παρακολούθηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αντίκτυπο στα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έγγραφο εργασία που είναι αποκλειστικά δικό μου δεν ετοιμάστηκε σε συνεργασία με άλλου και όδου εισηγητέ. Ο σκοπό λοιπόν αυτού του εγγράφου, εργασία είναι να υπάρχει μια συνολική παρουσίαση των ε, πληρέστων προγραμμάτων παρακολούθηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μια ε, απέτηση που εκφράστηκε τον περασμένο Ιούνιο εφόσον υπήρξαν σοβαρέ κατηγορίε. Υπάρχουν σχετικέ αντιδράσει και από Αμερικανικέ και Ευρωπαϊκέ Αρχέ σε σχέση με τα διάφορα προγράμματα και τον ερευνών για τις συγκέντρωση στοιχείων που έγιναν, συγκεντρώνοντα πόρου Αμερικανικού και Ευρωπαϊκού. Και οι Ηνωμένε και τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προηγμένε δυνατότητε υποκλοπή δεδομένων, ανάλυση και αποθηκευσή του. Όλα αυτά κατέστησαν εφικτά από το αυξημένη προσοχή που δόθηκε στι τεχνολογίε παρακολούθηση με προηγμένες μορφές υποκλοπής και γι' αυτό χρειαζόμαστε να διορθώσουμε τους αδύναμους μηχανισμούς παρακολούθησης που έχουμε. Το πιο σημαντικό είναι το εξή. Πολλά από αυτά τα βήματα πρόοδου έγιναν χωρίς να έχει προηγηθεί καμία δημόσια συζήτηση. Οι δικοί μας λοιπόν μηχανισμοί παρακολούθησης δεν έχουν προβληθεί το αυτοί σε δημόσιες διαβουλεύσεις. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε, το έγγραφο μάλλον επικεντρώνεται στο πλαίσιο διεθνώς και ευρωπαϊκός για τις υποκλοπές, τα προγράμματα παρακολούθησης που είχαν αντίκτυπο και στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα επικεντρώνομαι στα δεδομένα και τον ιδιωτικό βίο των ε, πολιτών και τα δικαιώματά τους, αλλά και το δικαίωμά τους να ασκήσουν προσφυγή, δικαίωμα σε ελεύθερη δίκη, δίκη και Ω προ το διεθνέ δίκαιο, σημασία έχει η κλίμακα και όγκο των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με τα προγράμματα μαζική παρακολούθηση, τα οποία αντικείται στο άρθρο 17 ε, του διεθνούς, της Διεθνούς Συμβάσεως του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της DCHR. Βάσει αυτών τα κράτη-μέλη εφόσον αναθέτουν στις εθνικές τους υπηρεσίες παρακολούθησης ε, ακόμα και τις, οποιαδήποτε δράση, ακόμα και τη συνεργασία με άλλες μυστικές υπηρεσίες άλλων κρατών μελών παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα ως προς τη δημοσιογραφία και τους ε, και όσους αποκαλύπτουν στοιχεία Εδώ έγιναν σχετικές έρευνες, όπως η έρευνα του Άλαν Westbridger, ο οποίος μίλησε για την αντίδραση κρατικών αρχών που ε, πολλές φορές είχαν αντίκτυπο σε ξένους πολίτες. Οι αποκαλύψεις του Σνόντεν που ένα αρνητικό αντίκτυπο στο κράτος και το πώς ε, επηρεάστηκαν οι δημοσιογράφοι από αυτό τον αντίκτυπο, αλλά και για τους ε, όσους αποκαλύπτουν στοιχεία, τους καταδότες εντό εισαγωγικών, και εκεί υπάρχει αντίκτυπος, αλλά πολλές φορές και τάση να κάνουν αντίπινα τα κράτη, να, προ... να προχωρούν σε αντίπεινα τα κράτη. Εδώ λοιπόν πρέπει να καλύψουμε και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα εκτό από την ελευθερία τη έκφραση και να συμβαστούμε και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο μαζί με άλλε οργανώσει των πολιτών όπω το Transparency International πρέπει να καλύψουν τις απαραίτητε υποχρεώσει σε σχέση με, το, με τους καταδότες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ανακεφαλαίωση των όσων λέει το σχέδιο εγγράφου εργασία που έχω ετοιμάσει και το οποίο μπορεί να δεχτεί τροπολογίες και βελτιώσεις. Για να προχωρήσουμε γρήγορα, Πρόεδρε, και να σεβαστούμε το χρονοδιαγραμμά, θα προχωρήσω αμέσω στην έκθεση τη Washington και μετά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ερωταπαντήσει. Θα προεδρεύσω ίσως αντικανονικά, κάπως αντιδημοκρατικά, αλλά για χάρη συντομία. Ε, για το έγγραφο της Washington, να πω ότι οι συνάδελφοι που ήταν μαζί γνωρίζουν ακριβώς τι έγινε. Τώρα, ε, έτσι για, την, ε, για τα πρακτικά, να πω επισήμως ότι ευχαριστώ τη γραμματεία, τον κύριο Άντουαν Κάιν και κάθε μέλος της γραμματείας της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά και τους συναδέλφους της ΑΘΕΤ, για μια επίσκεψη αντιπροσωπείας που ήταν λεπτομερέστατη και μας έδειξε τι κάνουν οι ομολόγοι μας στην Ουάσιγκτον. Πολύ δύσκολο να καταρτήσει κανείς ένα πρόγραμμα τόσο διεξοδικό και πλήρες όσο αυτό που ζήσαμε. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για αυτή την τόσο αποτελεσματική επίσκεψη που είχαμε. Τώρα δύο λεπτάκια για την ουσία. Είχα την αίσθηση ότι μέσα σε τρεις μέρες Ε, συζητήσαμε με ε, γερουσιαστές, με τον βουλευτή Ρότζερς, με την Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τις μυστικές υπηρεσίες, με την Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για το δικαστικό σύστημα και είχαμε επιτόπιες συναντήσεις χάρη και στην συμμετοχή της ΑΘΕΤ και είδαμε και τον επικεφαλής της NSA, την Κίθα Alexander, υπεύθυνος ασφαλείας είχαμε συναντήσεις με τα εποπτικά συμβούλια του βίου και της εμπιστευτικότητας για τις τεχνολογίες ασφάλειας τον Γενικό Γραμματέα Ρόμπερτ Λίντ τον Γενικό Πρέσβη για τα θέματα των μυστικών υπηρεσιών και στον Λευκό Οίκο τον Σύμβουλο του Αμερικανού Προέδρου θα ξεχάσω μια-δυο συναντήσεις, θα παραλείψω μάλλον μια-δυο συναντήσεις, αλλά στο τέλος είχαμε συνομιλίες με το εμπορικό επιμελητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα θέματα safe harbor, το ασφαλούς λιμένα. Ήταν πραγματικά πολύ ε, σφαιρική η εικόνα που σχηματίσαμε χάρη στις τόσο καλά οργανωμένες επισκέψεις. Και ένα δυο σχόλια τώρα. Αλήθεια είναι ότι Πολλά από αυτά που κάναμε στην Ουάσιγκτον μπορούσαμε να τα κάνουμε και εδώ, Ενδεχομένω. Αλλά θα συμφωνούν οι συνάδελφοι ότι άξιζε τον κόπο μέρο τη ερευνά μα να συμπεριλάβει και την Ουάσιγκτον, διότι υπάρχει υποστεθέμενη αξία εδώ για μα. Άνθρωποι που δεν θα είχαμε συναντήσει εδώ στι Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, ήταν άνθρωποι που συναντήσαμε εκεί, αλλά είχαμε και επαφέ με το Κογκρέσο. Νομίζω αυτές οι επαφές του Κογκρέσου ήταν και δρασματικές, Διότι για τα θέματα του RSA ήδη δημιουργήθηκε ένας πρώτος δεσμός και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και μετά από την έρευνα αυτή και την ολοκλήρωση της έκθεσης από το Κοινοβούλιο. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά πρόσφορο. Ένα παράδειγμα λοιπόν του γιατί αυτή η επίσκεψη ήταν ε, ιδιαίτερα χρήσιμη. Ένα μόνο παράδειγμα. Αυτά θα είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήταν αφοσιωμένοι και αφιέρωσαν χρόνο στο θέμα αυτό. Αυτές τις τόσο γεμάτες τρεις μέρες. Και απευθύνομαι και στο φανταστικό πρόεδρο που δεν κάθεται πλέον εδώ. Να προεδρεύσω. Ωραία λοιπόν, θα προεδρεύσω. Για τα έγγραφα εργασίας, <clears throat> νομίζω είναι γνωστά στους συναδελφούς. Να πάω στο επόμενο έγγραφο εργασία κατευθείαν. Καλά λοιπόν. Επόμενο έγγραφο εργασία. Εξωτερική πολιτική, πτυχέ εξωτερική πολιτική τη έρευνα για την ηλεκτρονική μαζική παρακολούθηση Ευρωπαίων πολιτών. Α, γύρισε ο πρόεδρο. Το έγγραφο αυτό το συντάξαμε εγώ και τρία μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η κυρία Αναγκόμες που είναι εδώ. Θα το σχολιάσει το έγγραφο, απλώς να κάνω και εγώ κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις και θα τις δώσω το λόγο. Εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Να πω αρχικά ότι ευχαριστώ την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και όσους από εκεί συμμετείχαν στην επίσκεψη της Washington ώστε να καταρτήσουμε αυτή την έκθεση. Το έγγραφο το κείμενο νομίζω δημιουργεί μια ε, συνολική σωστή ισορροπία μετά τις συζητήσεις της Επιτροπής ε, ΑΦΕΤ. Το βασικό σημείο ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης, η απόλυτη, απόλυτη εμπιστοσύνη στη σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτό ήταν το θέμα το βασικό. Το πλήγμα στην εμπιστοσύνη των σχέσεων μετά την μαζική παρακολούθηση πολιτών ήταν ένα μείζον ζήτημα που απασχόλησε του συναδέλφου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και αυτό σχολιάζουν στο έγγραφο. Πέραν των κατηγοριών για μαζική παρακολούθηση, το έγγραφο εργασία αναφέρεται και στι κατηγορίε κατασκοπία σε σχέση με του συνεργάτε τη κυρία Μέρκελ, το θέμα τρομοκρατία, τη τρομοκρατία και των εθνικών φορέων, και τη συνεργασία μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μιλά για την επίσκεψη τη αντιπροσωπεία στην Washington και κάποια άλλα τα βασικά σημεία. Νομίζω ήταν αυτά που αφορούσαν την ε, αυτά που σχολίασε και ο κύριο Άλπρετ για το πακέτο προστασία των δεδομένων. Νομίζω αυτό ήταν ένα σημαντικότατο σημείο που απασχόλησε την επίσκεψή μας στην Ουάσιγκτον. Δεν το ανέφερα προηγουμένως με αφορμή εκείνο τα το αναφέρω τώρα. Ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα των συναδέλφων και το ανέφερα και στην έκθεσή μα προ την ΑΦΕΤ. Η προσταθέμενη αξία της επίσκεψης της αντιπροσωπείας αυτής της έρευνας είναι ότι είμαστε οι μόνοι στο Ευρωκοινοβούλιο που διεξαγάμε έρευνα που ασχολείται ακριβώς με, έχει ως βασικό θέμα την προστασία των δεδομένων. Ακριβώς επειδή επιδιώκαμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη. Και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους τομείς του Safe Harbor, του ασφαλούς τομέα και αλλού, δεν θα έχουμε ποτέ σωστή διευθέτηση του θέματος των προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που είναι σημαντικό για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και σε ό,τι αφορά τι μυστικέ υπηρεσίε και την καταπολέμηση τη δημοκρατία. Θα ολοκληρώσω εδώ και, Πρόεδρε, να δώσω το λόγο, αν επιτρέπετε, στην κυρία Γκόμε, μια από τι του κειμένου τη Ευχαριστώ, Κλοντ. Και ευχαριστούμε για την εισήγηση, για τα σχόλια. που οποίο έκανε για το κοινό μας έργο θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σωστό το ότι πήγαμε μαζί και έτσι λοιπόν ε, είχαμε ε, επεξεργαστεί από δύο ε, οπτικές γωνίες από τα ΣΑΦΕΤ και από πλευράς ΛΥΜΠΕ και εγώ επίσης ε, δουλεύω και στην αντιπροσωπεία για τις είπα, πότε πάω τεχνικά στη Washington και ξέρετε ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν έχουν τόσο προσέξει αυτά τα οποία λέμε. Γιατί ακριβώς θεωρήσαμε ότι τώρα υπάρχει μεγάλη κρίση εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ ημών και εκείνων. Ε, γιατί βέβαια πέραν του φυσικά ε, σημαντικού αυτού ζητήματος ε, ήταν, το θέμα του τι θα γίνει κλπ. Δηλαδή, ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ομιλητές. Κογκρέσου, κυβέρνηση κλπ. Πολύ σημαντικές αυτές οι επαφές. Οπότε γι' αυτό και θεωρώ ότι τώρα αυτό διαμορφώσει την ανταπόκρισή τους Καταρχήν ήταν ε, αποδιοργανωμένοι, ανοργάνωτοι. Αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο Εξωτερικών, με την Υπηρεσία Ασφαλείας, Κίθα Αλεξάνδρ, με όλους αυτούς που σου μιλήσαμε τέλος πάντων. τελικά το Κογκρέσο στοιχήθηκε μάλλον με την κυβέρνηση. Συνειδητοποίησαν βέβαια ότι πρόκειται ακριβώς περί κρίσης εμπιστοσύνης και ότι η χρονική στιγμή ήταν μάλλον ατυχής γιατί έχουμε τώρα τις διαπραγματεύσει ε, για την εμπορική συμφωνία ή που θα καλύψει και τα ψηφιακά. Οπότε όλα τίθενται τώρα αμφιβόλα και γι' αυτό το λόγο και εμεί θεωρήσαμε και γράψαμε σε αυτή μας την έκθεση ότι εστιάζουμε την προσοχή μας ή την συμφωνία την προστασία των δεδομένων ε, ανεξαρτήτως της συμφωνία. συμφωνίας. Ακριβώς γιατί υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικέ επιπτώσει του ενός δημότος πάνω στο άλλο. Άλλο μεγάλο θέμα μεταξύ Κογκρέσου και κυβέρνησης είναι το ότι η βασική γραμμή του κυρίου Ρότζος έρχεται, ξέρετε, στις Βρυξέλλες. Οπότε αυτό είναι καλό στοιχείο ότι τώρα αυτό, αυτό βοηθάει τη ζήμωση και την συνόηση. Ότι τι να κάνουμε, το κάνουμε αυτό, αλλά το κάνουμε όλοι. Ποιος δεν το κάνει, το κάνει η Γαλλία, το κάνουν όλοι. Οπότε σιγά, σιγά την υπόθεση, σιγά την προστασία. Όμως, ο Γιωτσέτης Φανιστάιν δεν είπε το ίδιο, γιατί μιλήσαμε και με τη Σχετική Επιτροπή της Γερουσίας και όποτε ήταν πάρα πολύ βασικό το ότι όχι μόνο έγινε αυτή η συνάντηση της, της Γερουσίας με μας και με τον Κίθα Αλεξάνδερ, αλλά τα είπε και δημοσία και επέκρινε την υπηρεσία ασφαλείας, την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας για όσα έγιναν. σε σχέση και με τη γραμμή που ετήρησε η κυβέρνηση. Οπότε, έτσι. Ε, ξεκίνησε μια λυσιδεντή δράσεων, είχαμε την ε, συνέντευξη τύπου, εκεί η Αλεξανδρή και άλλοι αποφασίσαν ότι τώρα που τα είπε αυτά η στην βγήκε και είπε τέτοια πράγματα Ανεγνώρισε ότι έγινε κάτι στραβό. Δεν απέδωσαν οι δικαστικές και άλλες εγγύσεις. Οπότε αυτό τους κινητοποίησε. Χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου, ο συναγερμός. Και γίνανε πιο επιθετικοί οι στρατηγικοί τους. Οπότε παγίως όσον αφορά την κυβέρνηση συνομιλούμε με την ε, με τους συμβούλους του Ομπάμα, με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπά Και αυτή τη φορά αναγνώρισαν ότι κάτι έγινε στραβά, κάτι πήγε στραβά και ε, ξέρετε, μου τον Ομπάμα ασφαλεία είπανε ότι να το συζητήσουμε, να αντλήσουμε συμπεράσματα, να μάθουμε κάτι από αυτά. Και να δούμε πώς θα βελτιθεί η κατάσταση. Αυτό ήταν ε, το καλό, το θετικό. Αυτό που ήταν όμως το αρνητικό είναι ότι στο State Department, κυρία Γκόμες λέει ο πρόεδρος, κάποιοι βουλευτές θεωρούν ότι πιέζει ο χρόνος, οπότε αν μπορείτε συνοψίσατε. Πέστε μας για την έκθεση, γιατί πέραν τα, των του ταξιδίου. Οπότε τώρα η ένδικη προσφυγή, η η να λύση του ζητήματος που είναι σημαντικό για μας ε, δεν προβλέπεται στην Αμερική βέβαια εκεί ε, ε, έχουν έχουν, έχουν διεθνείς δεσμεύσεις και είπαμε ότι άμα κάνουμε εσάς τη χάρη θα έρθουν και οι Αφγανοί να ζητήσουν τα ίδια, έτσι λέγανε. Όμως, πιστεύω θα πρέπει να μείνουν στα αιτήματά μας χτυπήσουμε το χέρι. Και η Επίτροπος Ρέντε πριν από μια δύο μέρες είπε ότι τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει και αυτά να περιληφθούν στι διαπραγματεύσει, αλλά είναι αδιαπραγμάτευτα τα δικαιώματα. Ναι, αδιαπραγμάτευτα, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε εγγύσει για τα δικαιώματα των ε, πολιτών μα και να ωφεληθούν και οι Αμερικανοί πολίτε Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ελάχιστο πρότυπο, ελάχιστο στάνταρ επίπεδο τέλο πάντων κάποιου είδου δυνατότητα ε, προσφυγή στη δικαιοσύνη και να μην υπάρχουν ορισμένε διακρίσει ακριβώ όπω ισχύει τώρα εδώ, αλλά και στην Αμερική. Αυτό τι δείχνει, ότι χρειάζεται εποπτεία, χρειάζεται άσκηση δημοκρατικού ελέγχου και ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Άλλωστε ξέρετε ότι υπάρχει κατάτμιση των αρμοδιοτήτων. Άλλα γίνονται σε εθνικό επίπεδο και άλλα γίνονται σε εθνικό <coughs> όσον αφορά την εθνική ασφάλεια. Κύριε Γκόμε, σα ευχαριστούμε. Κλοντ, η σκητάλη ξανά ει εμά. Ναι, κοιτάξτε τώρα, επειδή έχει περάσει και η ώρα, α τελειώνουμε, κύριε Πρόεδρε. Ας περάσουμε στην παρουσίαση του εγγράφου εργασίας ε, για την δημοκρατική εποπτεία. Ε, νομίζω μπορεί να κάνει την εισαγωγή η κυρία Ίνετφελντ. Σοφή, με συγχωρείς, ε, με συγχωρείτε, η κυρία Μάνστρομ. ε, ότι καθυστερήσαμε, ζητώ συγγνώμη από αυτήν και το προσωπικό της. Μπορούμε νομίζω να συνεχίσουμε. Κοιτάξτε μα, η συζήτηση αυτή είχε προγραμματιστεί 16 και 40. Οπότε έχει πάει 5 ώρα ήδη, έτσι. Αλλά τι να πω, δεν είναι και το τέλος του κόσμου ότι, ότι καθυστερήσαμε τόσο πολύ. 20 λεπτάκια καθυστέρηση δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ε, ναι, κοιτάξτε, στο κοινοβούλιο με, με χρόνους κοινοβουλίου δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά άμα σκεφτούμε ότι είναι και πέμπτη απόγευμα, Κοιτάξτε από δημοκρατική σκοπιά να πω. Γιατί δεν είναι εδώ και η κυρία Ένστ. Δεν ξέρω, είναι και η βοηθός της εδώ πέρα. Να συνεχίσουμε χωρίς αυτήν. Σόφι, εσείς τι λέτε. Ε, είστε και εσείς ε, συνεισηγήτρια. Θέλετε να εξηγήσετε κάποια πράγματα. Είναι έκθεση του κυρίου Μωραές, ε, της κυρίας Σίνετφέλντ και της κυρίας Ένστ. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω την εισαγωγή, αλλά θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όλοι νομίζω συμφωνούν πως η εποπτεία των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών είναι ένα ζήτημα κλειδί που προέκυψε. Και αυτό διδαχτήκαμε από όλες τις αποκαλύψεις των ΜΜΕ είναι πως θα πρέπει να ξεκινήσει η εποπτεία στο εθνικό επίπεδο ε, όπου αποτυγχάνει. Έτσι. Είναι αδύναμη και πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών. Και βλέπουμε πως υπάρχει περισσότερη συνεργασία, νέες τεχνολογίες ε, που τους δίνουν δυνατότητα περισσότερη συνεργασία και είναι βασική αρχή σε οποιαδήποτε φιλελεύθερη δημοκρατία πως ε, κάθε εξουσία πρέπει να ελέγχεται. Έτσι. Οπότε μια βασική σύσταση πρέπει να είναι πως τα εθνικά συστήματα δημοκρατικής εποπτείας επί των μυστικών υπηρεσιών πρέπει να ενισχυθούν και εάν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να το κάνουν λογικό θα ήταν να γίνει επί τη βάση των ιδίων προδιαγραφών. Γιατί αν συνεργάζονται οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε σε συστήματα εποπτείας σε άλλα κράτη-μέλη. για να γίνονται σεβαστά με τον ίδιο τρόπο τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίας ε, και να μην υπάρχει πρόβλημα μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας. Δεύτερον, έχουμε εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της μυστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επισήμως δεν υπάρχει, δεν έχει καν βάση στις συνθήκες νομίζω πως συμπεριλαμβάνεται στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, με μια, με, με μια διακεκομένη γραμμή. Αλλά ε, υπολογίζεται πως υπάρχουν ήδη 72 με 100 άτομα που εργάζονται. Ε, μυστική μυστική υπηρεσία. Αλλά υπάρχει. Αλλά νομίζω πως πρέπει να... Ε, δούμε τι γίνεται με την Incent αλλά και να δούμε με τι γίνεται με τις συνορικές δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν υπάρχουν στο έγγραφο εργασίας. Και τι άλλο έχουμε τώρα, εδώ πέρα ερωτήσεις για συζήτηση που θα γίνουν τελικά συστάσεις. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω τέταρτη παραγραφό στον τίτλο «Λύσεις». Λέει, ομάδα εργασίας πρέπει να συσταθεί. Εγώ ανατριχιάζω όταν τα ακούω αυτά τα πράγματα. Ομάδα υψηλού επίπεδου, ομάδα εργασίας, task force κτλ. Ξέρετε, παραπέμπονται έτσι τα θέματα στις ε, καλένδες. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να το δούμε γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου. Θα υιοθετήσουμε τις συστάσεις πριν ακριβώς λήξει και πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός, ένας τρόπος να διασφαλίσουμε πως το Κοινοβούλιο αμέσω μετά τις εκλογές θα συνεχίσει το έργο αυτό και πως οι συστάσεις θα υιοθετηθούν. Τώρα, αν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι καλύτερο από το ομάδα υψηλού επίπεδου, ευχαριστώ. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να φροντίσουμε ε, ώστε ε, τα συμπεράσματά μας να μην καταλήξουν σε κάποιο σιρτάρι σαν αυτά του Έσελον, αλλά να γίνει κάτι παραπάνω. Όχι μόνο να λέμε ναι, ναι, πρέπει να συνεχιστεί το έργο αυτό κτλ να, ναι. δοθεί μια συνέχεια. Μια τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Διαφάνεια, γιατί μιλάμε για διαφάνεια και δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα να είναι κατά της διαφάνειας. Ταυτόχρονα υπάρχει και κανονισμός διαφάνειας ο οποίος όμως ε, δεν είναι πολύ ισχυρός. Ειδικά το Συμβούλιο δεν το εφαρμόζει πλήρως. Ε, ξέρω πολύ καλά τι λέω από πρώτο χέρι γιατί έχω ζητήσει πάρα πολλά έγγραφα και κάποια από τα αιτήματα, μάλλον οι απορρίψεις της ε, Κομισιόν κατέληξαν και στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Όμως οι προτάσεις για να αναβαθμιστεί ο κανονισμός έχουν κολλήσει κάπου, έτσι. Και πρέπει εδώ πέρα να είμαστε ανυποχώρητοι πως οποιαδήποτε αναθεώρηση του κανονισμού πρέπει να οδηγήσει σε ενδυνάμωσή του, έτσι. Οπότε ανησυχώ για φήμες που ακούω ότι κάποιες ομάδες εντός του Κοινοβουλίου θέλουν να προτείνουν κατά βάση ε, να δεχτούμε ό,τι μας προτείνει το Συμβούλιο και η Κομισιόν και να έχουμε έναν εξασθενισμένο τέτοιο κανονισμό. Εγώ είμαι εναντίον. Και τέλος, κάτι το οποίο είχα προτείνει στην έκθεση μου, στην ετήσια έκθεση διαφάνειας, έχουμε κανόνα, αλλά δεν έχουμε διαδικασία για την κατάταξη των εγγράφων. Οπότε, εάν κάποιος μας αρνηθεί την πρόσβαση. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή μόνο στο δικαστήριο μπορούν να πάνε οι πολίτες. Εγώ βήμαι στα δικαστήρια 5-6 χρόνια. Το κόστος είναι απαγορευτικό για το μέσο πολίτη. Οπότε χρειάζονται δικασίες για την κατάταξη των εγγράφων. Αυτό το οποίο λέμε βαθμός ασφαλείας στα ελληνικά. και επίσης ένας ε, φορέας εποπτείας, ε, ε, κάποιος ο οποίος θα είναι υπεύθυνο για τη διαφάνεια, έτσι, για να εφαρμοστούν επιτέλους αυτές οι συστάσεις που κάνουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Ενετφέλντ, ευχαριστώ. Κλοντ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή στο κείμενο. Δεν θέλω να χασομερίσουμε παραπάνω. Απλώς μια ένα σχόλιο. Ότι η υποπτία απαιτεί κρατική ε, ευθύνη και νομική αρμοδιότητα σε επίπεδο φορέων των κρατών μελών, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε να δούμε και στο κείμενο, πώς ακριβώς θα υπάρξει ευρωπαϊκή εντολή για τα θέματα αυτά και ακριβώς θα δούμε τι συστάσεις μπορούμε να κάνουμε. Λόγω χάρη κάποιες συστάσεις για την ενίσα και για τους πολίτες ιδίω προ όφελο των πολιτών όπου υπήρξε συνεργασία μεταξύ μυστικών υπηρεσιών. Θέλω να το τονίσω αυτό γιατί είναι σαφέ ότι πρέπει να κάνουμε συστάσει και για αυτά που γίνονται από του ε, εθνικού ερευνητέ. Πρέπει να υπάρχουν διαθετήσει διαφάνεια για τι εθνικέ μυστικέ υπηρεσίε. Αλλά εφόσον δεν έχουμε εμεί αρμοδιότητα, θα πρέπει να το ζητήσουμε από τι εθνικέ αρχέ. Πρέπει να είμαστε αρκετά τολμηροί και να φανούμε αποφασιστικοί, να το απαιτήσουμε και να μην ε, επεκτηθούμε των ευθυνών μας, γιατί και εμείς εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Να προσθέσω λοιπόν και εγώ αυτό το σχόλιο στα υπόλοιπα που είπατε. Πολύ καλή παρουσίαση των γραφών Εργασίας. Θα έλεγα το ίδιο ακριβώ. Τίποτα δεν πρέπει να μας σταματήσει από το να διατυπώσουμε συστάσεις. Δεν μιλάμε για επικουρικότητα ή αρμοδιότητε Ευρώπη ή όχι, μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να γίνουν συστάσει. Εάν οι εθνικέ κυβερνήσει επιλέξουν να τι αρνοήσουν, τότε να εξηγήσουν αυτοί στου πολίτε του γιατί δεν θέλουν εποπτεία. Εμεί όμω πρέπει να το κάνουμε και να εκπληρώσουμε το καθήκον μα προ του πολίτε. Να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Θε το λόγο, θε να καθυστερήσουμε εδώ. Θα σου δίνω το λόγο για το επόμενο. Το ξέρω, αλλά πριν πάρω το λόγο για το επόμενο έγγραφο εργασία, θέλω να παρέμβω και να πω ότι απολύτω συμφωνώ. Θα ήθελα να αναφερθεί η η εξή ιδέα. Μιλάμε για ένα όργανο αποπτία της Europol. σω αυτό θα μπορούσε να συμπεριλάβει την Ίντσεν και την υπόλοιπη ομάδα των μυστικών υπηρεσιών. Θυμηθείτε, και εγώ είχα εκπλαγεί όταν άκουσα ότι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν 4-5 μέλη που ασχολούνται με την υποπτία της Δεν το ξέρατε, υπάρχουν. Είναι η διαθεσμική συμφωνία με το Συμβούλιο. Με τα κάτι μέλη όμως μόνο. Εγώ το βλέπω γελίο να με γνωρίζουμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αξιολόγηση του πώς γίνονται σεβαστά και το καθεξής και για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι γελίο να μην έχουμε γνώση. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι συνάδελφοι αυτοί προφανώς δεν αισθάνονται υποχρεωμένοι να μας ενημερώσουν, να έρθουν σε επαφή μαζί μα. Βρίσκω ότι υπάρχει ένα, σαφό κενό, ένα σαφές κενό επικοινωνίας εδώ. Η θεσμική συμφωνία αναφέρει ότι μόνο οι δύο μεγαλύτερες ομάδες θα λαμβάνουν ενημέρωση. Τι να πω, δεν ξέρω. Ποιοι θα είναι αυτοί, το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι μαζί. Κανείς εδώ δεν φαίνεται να γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν σας το λέω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση και με ενοχλεί πάρα πολύ. Πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους. Κυρία Γκόμες, ε, διευκρινίστε το. Εκτός μικροφώνου κυρία Γκόμες. Πώς θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Ξέρω ότι υπάρχει και θα έπρεπε να συμμετέσχουν τουλάχιστον οι συντονιστές του Γεδομένου Προεδρείου της ΑΦΕΤ. Ένας από τους, ως, μίας, ως μία από τις εισηγητρίες το ζήτησα και εγώ. Αλλά η απάντηση δεν έφτασε ακόμα. Δεν έχω συμμετάσχει λοιπόν ακόμη καθόλου στην όλη διαδικασία. Δεν γνωρίζω. Ό,τι για να έχει γίνει δεν με αφορά ω συντονίστρια, λέει η κυρία Γκόμε, πρόεδρο. Θέλετε το λόγο. Ε, θα ρωτήσω ε, ε, γι' αυτό τον πρόεδρό μας την ΑΦΕΤ, τον κύριο Μπρόκ. Ναι, ναι, νομίζω θα πρέπει να γίνει κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό. Όχι, δεν είναι υπηρεσία πληροφοριών. Ε, είναι κέντρο συλλογής και αναλύσεως ε, στοιχείων ε, και πληροφοριών που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και ενεργεί ως σύμβουλος προς την υπηρεσία ε, εξωτερικής δράσης. Ξεκίνησε επί Σολάνα και τώρα βοηθά την κυρία Άστον. Δεν είναι υπηρεσία πληροφοριών. Συλλογή πληροφοριών. Αναλύει, αναλύει πληροφορίες. Δεν συλλέγει. Μα αυτό κάνουν όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών, λέει ο κύριος Άλμπριχτ. Λέγεται Ίνσεν. Δεν υπάρχει νομική βάση σχετική και ούτε ασκείται κανένα έλεγχο, ούτε ξέρουμε τι, τι, γίνεται εκεί. Πρόεδρο. Τώρα μόλι το έμαθα. Δεν το είχα υπόψη μου. Δεν ήξερα ότι αυτό είναι θέμα της ΑΦΕΤ, εγώ τώρα προσπαθώ. Προσπαθώ να ενημερωθώ από τους συνεργάτες μας, τις υπηρεσίες μας, τη γραμματεία μας και αν μου επιτρέπετε να σα πω τι μου έγραψαν. Just to let you know that the current interinstitutional agreement on transmission of confidential information είναι εμπιστευτικέ πληροφορίε, λέει ο πρόεδρο. They only only deals for foreign affairs AFET, but there is ε, ξεκίνησε αυτό για την άφετα, όμως υπάρχει μια γενοργία εκδοχή και αφορά και θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών, οπότε και η ΛΥΜΠΕ θα είναι συναρμοδία το μέλλον για αυτό. Πρόκειται για αυτή την συμφωνία της ε, τόρης διαβίβασης εμπιστευτικών πληροφοριών και βέβαια ξεκίνησε ως θέμα της ΑΦΕΤ, οπότε προς ενημέρωσή σας. Σας τα είπαμε όλα αυτά για τις επιφυλάξεις Οπότε Πάμε τώρα για το τι γίνεται με αυτή την παρακολούθηση και τα όσα προβλέπονται για τους ασυνδεδομένων. Αυτό είναι μια έκθεση του κυρίου Μωράς και του κυρίου Άλμπρεχτ. Τώρα, ποιο ημών θα ήθελε να κάνει την εισήγηση. Κύριε Άλμπρεχτ, έχετε το λόγο. Πόσα λεφτά θέλετε να μιλήσω, Πόσα θέλετε. Ε, αφήστε λίγο χρόνο για να για απαντήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Καλά, καλά. Απλώς ήθελα να ξέρω. Καλά, σε δύο και θα σας τα πω. Κοιτάξτε, έχουμε αυτό το έγγραφο εργασία, το οποίο αφορά αυτές τις παρακολουθήσεις, υποκλοπές και έτσι για να θυμηθούμε περί τίνος ε, συζητούμε και την άλλη μεριά έχουμε το τι γίνεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπα και την άλλη μεριά τι γίνεται με το πρωτογενές ε, κοινωνικό δίκαιο και το δίκαιο προστασία δεδομένων. Και καταλήξαμε στο ότι γενικά τα κρατημέλη υποχρεούνται να τηρούν, να συμμορφώνονται προς το πρωτογενές και το δευτερογενές κοινωνικό δίκαιο. Παρακαλώ, κλείνετε το μικρόφωνο σας γιατί έχει παρεμβολή, δημιουργεί παρεμβολή. Οπότε έχουμε το δίκαιο προστασίας δεδομένων και τα σχετικά με το κυβερνό έγκλημα. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά επίσης υπάρχει το θέμα της εθνικής ασφαλείας που είναι μια εξαίρεση που κατησχύει τέλος πάντων των άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, οπότε και συνεχίζεται η προβληματική για αυτήν την εξαίρεση της εθνικής ασφαλείας. Οπότε και να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν αυτά τα μέτρα παρακολούθησης να μην διέπονται από τις διατάξεις του δικαίου που είπαμε. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ κατά. Όμω είπαμε ότι οι διατάξει λίγο των δεδομένων ε, δεν σχετίζονται, δεν θα έπρεπε να υπάγονται στι διατάξεις για την εθνική ασφάλεια. Όποτε έχουμε την εθνική ασφάλεια των ε, τρίτων χωρών που δεν δημιουργεί εξαίρεση ε, από τις διατάξεις του κοινωτικού δικαίου. Άρα εξαίρεση χωρί μόνο για τις δραστηριότητες που αφορούν την εθνική ασφάλεια των κρατών μελών. Και θα πρέπει με το πρωτογενές και το δευτερογενές δίκαιο να ξεκαθαριστεί ακριβώς πώς οριοθετείται η έννοια της εθνικής ασφαλείας. Επίσης να ξεκαθαριστεί για τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων, πώς θα έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εφαρμογή. Και ότι τα μέτρα τα οποία προβλέπονται δεν παραβιάζουν το κοινωτικό δίκαιο. Δεν αποτελούν παραθυράκια δηλαδή, στην ισχυρή ρύθμιση. Και δεν παρακάμπτουν το νόμο. Επίσης, έχουμε τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια της αστυνομικής και διοικητικής συνεργασίας. Εδώ είναι θέμα εφαρμογής του δικαίου και όχι α, θέμα εθνικής ασφαλείας. Να δούμε πώς θα θωρακιστεί η προστασία των δεδομένων για τις δραστηριότητες που αφορούν τα κράτη-μέλη αλλά και τρίτα κράτη-μέλη. Τέλος δε, θα πρέπει ο κανονισμός να λέει ότι αν κάποιος αποσπάσει κάποια δεδομένα ε, όπως προβλέπει το άρθρο 6 κατά παραβίαση των κειμένων διατάξεων δεν θα λαμβάνουν υπόψη αυτά τα δεδομένα σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε εδώ πέρα μια σειρά συμπερασμάτων στο κείμενό μας, αλλά δεν θα σας πω τίποτε άλλο, θα σταματήσω εδώ. Δεν θέλει κάποιος να λέει το λόγο, οπότε προχωρούμε. Πάμε στο επόμενο σημείο, λέει ο Οπότε... Τώρα, έχουμε το τρίτο τελικό τμήμα της συστήσεως που είναι οι επιπτώσεις των ε, μαζικών παρακολουθήσεων και αποκλοπών όσον αφορά την παραβίαση των εμπιστευτικών σχέσεων συνηγόρου πελάτου. Τώρα μπήκαμε στα πιο εξειδικευμένα γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρόκειται να μας το εξηγήσουν. Να το... Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. τιμή μας που ήρθατε θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Jonathan Goldsmith, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της νόσεως του Φορέα, τέλο πάντων των Δικαιωρικών Συλλόγων και Νομικών Συλλόγων της Ευρώπης. Και ε, ο φορέας των προεδρικών τον Οκτώβριο προέβη μια ανακοίνωση σε σχέση με τις συνέπειες αυτών των παρακολουθήσεων και υποκλοπών. Αφορά το επαγγελματικό απόρριτο του δικαιωρικού επαγγέλματος, το κράτο δικαίου στην Ευρώπη κλπ. κλπ. Επομένω, είσαστε ο πιο κατάλληλο για να μα τα εξηγήσετε όλα αυτά. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ. Ε, περιμένω λίγο τις διαφάνειες κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ετοιμάζονται τώρα. Έτοιμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή που προσεκάλεσε την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης. Ε, τα μέλη μας είναι δικηγορικοί σύλλογοι. Αντιλαμβάνεστε. Α, ωραία. Είναι το ο χάρτης, αλλά δεν μπορείτε να τον δείτε. Δείχνει ποια είναι τα μέλη μας. 32 πλήρη μέλη έχουμε, 12 μέλη παρατηρητές και εκπροσωπούμε πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους δικηγόρους. Και βεβαίως, ε, όπως είπατε, πράγματι βγάλαμε μια δήλωση για τον αντίκτυπο που, έχει, ε, που έχουν αποκαλύψει ο κ. Σνόντεν στο επαγγελματικό απόρριτο. Το βασικό ερώτημα μπορεί να τεθεί πάρα πολύ απλά. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που θα θέλαμε να θέσουμε είναι το εξής. Έστω ότι εγώ είμαι ο δικηγόρος του Σνόντεν. Τι εγγυήσει έχω για το απόρριτο μεταξύ εμού και του κυρίου Σνόντεν. Ξέρουμε ήδη την απάντηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια εγγύηση για το επαγγελματικό απόρριτο μεταξύ μας. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Πρέπει να σκεφτούμε κάνα δύο λεπτά το τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει επαγγελματικό απόρριτο. Μιλάμε λοιπόν για επαγγελματικό απόρριτο πελάτη δικηγόρου. Ισχύει σε όλα τα κρατη έχει διαφορετικά ονόματα, κατ' ουσίαν ε, είναι ε, το ίδιο πράγμα εγώ θα το πω επαγγελματικό απόρριτο, αυτό κατ' ουσίαν προστατεύεται από τους νόμους, τα συντάγματα ή τον ποινικό κώδικα της κάθε χώρας. Αναγνωρίζεται σε κάθε κράτος μέλος, αλλά και επανειλημμένα στην ομολογία του ΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολλά πράγματα λοιπόν μπορούμε να πούμε. Πρώτον, παρά το ότι εμεί το λέμε επαγγελματικό απόρριτο, κάποιοι άλλοι το λένε προνόμιο, ε, δεν είναι το νόημα να ωφεληθούν οι πολίτες, αλλά οι πελάτες, αλλά οι πολίτες, με συγχωρείτε. Για να ε, προστατευτούν βεβαίως πρώτα απ' όλα οι πελάτες και να υπάρξει ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό. Οι πελάτες πρέπει να μπορούν να μιλάνε με τον δικηγόρο τους, να του πούν την αλήθεια και ε, βεβαίως υπό μυστικότητας. Μπορεί να φοβούνται, μπορεί να έχουν κάποια πράγματα που θα τους εκθέσουν. Άλλες παρανομίες που θέλουν να κρύψουν. Παρ' όλα αυτά είναι προ το συμφέρον γενικά της απονομή της δικαιοσύνης Α, εμπιστεύονται πλήρως τους δικηγόρους τους οι πελάτες, αυτό είναι προς το συμφέρον τους και προς το συλλογικό μας συμφέρον. Έτσι ε, προστατεύεται, μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιλογές που μπορεί να μην γνωρίζει ο πελάτης ε, μέχρι να αποκαλύψει όλη την αλήθεια στον δικηγόρο του. Οπότε όπως σας είπα βοηθάει και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί, να σας δώσω ένα παράδειγμα πρέπει να υπάρχει εάν θέλετε μεταξύ των μερών μια κάποια ισοτιμία. Και σαφώς, εάν μία πλευρά διαβάζει όλα τα μηνύματα και την αλληλογραφία και η άλλη δεν το ξέρει, βεβαίως δεν υπάρχει κάποια ισοτιμία. Η πλευρά η οποία διαβάζει, είπαμε, όλα τα μηνύματα μπορεί καλύτερα, αν κάνει ε, και άλλες παρανομίες, ε, να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε πρέπει να υπάρχει αυτή η ισοτιμία και το επαγγελματικό αυτό απόρριτο που υπάρχει, υπάρχει ακριβώς για να υπάρχει ορθή απονομή της δικαιοσύνη. Πρέπει να σου πω πως δεν υπάρχει για κάποιο άτομο μπορεί να πει κανείς ε, γιατί ο κύριος Σνόουντεν να έχει αυτό το πλεονέκτημα όταν ε, ε, φρόντισε ο ίδιος να αποκαλύψει τα μυστικά των πάντων. Και τώρα λέει «Α, εγώ έχω απόρριτο». Μα ε, το θέμα δεν είναι ο κύριος Σνόντεν, έτσι, υπάρχει για όλους εμάς, για τους πολίτες, για το κοινό καλό. Και γι' αυτό τον λόγο, εξαρτήτως του πόσο ε, βαρύ μπορεί να είναι το έγκλημα, ε, συνήθως ε, το μέτρο του πολιτισμού μας είναι πως όσο πιο βαρύ το έγκλημα, τόσο πιο ορθή πρέπει να είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Και υπάρχει αυτό σε διάφορα σε διάφορους τομείς του δικαίου και στο ποινικό δίκαιο και στο αστικό έτσι η περίπτωση Snowden είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η κατασκοπία επηρεάζει και το αστικό τμήμα της υπόθεσης γιατί δεν είναι μόνο για εγκλήματα αλλά και για εμπορικά μυστικά έτσι εμπορικά μυστικά εταιριών που ε, Μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο κατασκοπίας ε, και σαφώς είναι προς το συμφέρον των κρατών σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν πρόσβαση σε εμπορικά μυστικά π.χ. τεχνολογικά μυστικά στην περίπτωση που κάποιος αναπτύσσει μια τεχνολογία που θα αφορά την κατασκοπία. Στρατιωτικά μυστικά, γενικά εμπορικά μυστικά που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες ξένες εταιρείες ε, να έχουν ένα μειονέκτημα. Αυτά περνάνε από τα δικηγορικά γραφεία Μία ανησυχία είναι μάλιστα πως ε, το δικηγορικό γραφείο είναι ο αδύναμος κρίκος στην όλη αυτή την υπόθεση, γιατί όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν τα μέτρα τους και πρέπει να φροντίσουμε το ίδιο να κάνουν και οι δικηγόροι. Οπότε, αυτή είναι η βάση, όπως είπα, του επαγγελματικού απορρίτου. Ποια είναι η σχέση λοιπόν μεταξύ επαγγελματικού απορρίτου και δημοκρατίας που μας απασχολεί. Κατ' ουσίαν ε, η δημοκρατία βεβαίως ε, σημαίνει πως ε, μπορεί κανείς να ψηφίζει, αλλά όπως ξέρουμε και από το Ιράκ και τα λοιπά, αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Κοινωνία των πολιτών και κάποιους μηχανισμούς και ένας από τους μηχανισμούς αυτούς, στους οποίους βασίζεται η δημοκρατία, είναι η δυνατότητα να διορθώνει τα λάθη της που την διακρίνει από τις δικτατορίες, όπου βεβαίω είναι δύσκολο να αλλάξει ο δικτάτορας ή να αλλάξει μια κατάσταση. Και βέβαια προσπαθούμε να αποφύγουμε τα λάθη αυτά. Προφανές παράδειγμα το κοινοβούλιο. Ε, μην ξεχνάτε ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο πως ε, η αντιπολίτευση είναι η ε, πιστή αντιπολίτευση της ε, αυτής ε, έτσι, δηλαδή είναι πιστή ενώ στο κράτος, αλλά αντίθετη με την κυβέρνηση. Και μην ξεχνάμε πως ε, εάν δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο υπάρχουν τα δικαστήρια και οι δικηγόροι. Μια άλλη επίσης ε, σημαντική εξουσία. Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα ε, η υπόθεση με τον Μέρντοχο που κοινοβούλιο κυβέρνηση και ο τύπος ε, ήταν υπό το καθώς εκφοβισμού από τον Μέρντοχ στις περίπτωση στην οποία προσπάθησαν να αποκαλύψουν κάποιες ε, λανθασμένες πρακτικές. Εκεί πέρα τα δικαστήρια έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να αποκαλύψουν ε, κάποια στοιχεία. Ακόμα και τα θύματα διασημότητες ε, φοβόντουσαν. Το μόνο, μόνος τρόπος λοιπόν είναι να διορθωθούν. Ο μόνος τρόπος να διορθωθούν αυτά τα λάθη είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στον δικηγόρο και να μην ε, είναι διαθέσιμα τα ε, μυστικά αυτά σε όποιον μπορεί να υποκλέψει. Το θέμα λοιπόν είναι τι σημαίνουν αυτές οι μαζικές παρακολουθήσεις για τις σχέσεις ε, πελάτη δικηγόρου. Έχει φύγει, ε, όπως σας είπα και απέδειξα, νομίζω ένα βασικό στατικό στοιχείο της δημοκρατίας ε, και του κράτους δικαίου. Έτσι. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, το κράτος έχει πρόσβαση στα πάντα, ακόμα και στην εμπιστευτική επικοινωνία δικηγόρου με τον πελάτη. Και βεβαίως ε, βλέπουμε πως έχει υπάρξει συχνά και από τους πράκτορες ε, κατάχρηση αυτών των δεδομένων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δεδομένα, υπάρχει χρήση και κατάχρηση. Όπως σας είπα, ανησυχούν πάρα πολύ. Δεν φαίνεται να υπάρχει επίση κάποια λύση. Εμείς ε, ως ε, Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης δεν ξέρουμε τι να πούμε στα μέλη μας για να πούν και αυτοί στα μέλη τους του δικηγόρους για την ασφάλεια των επικοινωνιών. Δεν υπάρχει τεχνολογία από όσο ξέρουμε που να μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε μέχρι να λυθεί αυτό το ζήτημα συνειδητοποιούμε πως ε, σημαντικό κομμάτι της δεοντολογίας ε, των δικηγόρων έχει μόλις ακυρωθεί. Και αυτό, όπως είπα, έχει μεγάλη σημασία γιατί επηρεάζει τους πολίτες. Οι συστάσεις μας, λοιπόν, χωρίζονται σε νομικές και τεχνικές λύσεις. Τι θέλουμε λοιπόν να δούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο προστασία του επαγγελματικού απορρίτου από την παρακολούθηση, την κρατική. Έτσι, προφανώς, για προφανείς λόγους, τα μέλη μας στο εθνικό επίπεδο ανησυχούν. Γιατί βέβαια πρέπει να αντιδράσουν και έχουν απέναντι τις κυβερνήσεις τους. Έτσι. Εντάξει, και τους λένε πως η κατασκοπία είναι καλό πράγμα, μας προστατεύει αλλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο ακούμε πως είτε δεν υπάρχει υπηρεσία κατασκοπίας, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να θέσει κάποιες προδιαγραφές. Γνωρίζω πως η εθνική ασφάλεια δεν είναι βεβαίως ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε χρειάζεται κάποια προστασία στο επίπεδο αυτό. Θέλουμε λοιπόν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και ε, για λόγους εθνικής ασφαλείας. Όσον αφορά τις τεχνολογικές λύσεις, θα θέλαμε κάποιες εγγυήσεις πως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ε, και όλα αυτά θα ε, σέβονται την, το επαγγελματικό απόρριτο. Σας ευχαριστώ. Goldsmith, not bad. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Goldsmith και σας ευχαριστούμε μια που μας παραδώσατε εδώ πέρα μαθήματα συνευματικού δικαίου που ε, από δικού σας στόματος είναι κάτι πάρα πολύ αξιόλογο μια που εκπροσωπείται τους δικηγορούς λόγους όλες της Ευρώπης. Έτσι έχω την αίσθηση ότι ακούσαμε πολύ περισσότερα από όσα θα ε, μας λέγατε θεωρητικά όσον αφορά δηλαδή το θέμα μας δηλαδή όσον αφορά τη σχέση εμπιστοσύνη αυτό δεν ήταν η κίτρινη κάρτα στις παρακολουθήσεις που βγάλατε. Ήταν ε, ένας ε, συναγερμός πραγματικός, όπως μας τα είπα. Και τώρα, ο εισηγητής και οι εισηγητές για ερωταπαντήσεις. Ερωταπαντήσεις όλα μαζί, Πρόεδρε. Ναι, ναι, σημαντικό αυτό που με τη συζήτηση. Σημαντικές σχέσεις ε, πελάτ και όσα μας είπατε. Και μας τα είπατε ξεκάθαρα. Και βέβαια μπορούμε να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. πήγαμε και στην Washington στα πλαίσια τη έρευνα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό το οποίο διέρευσε, δηλαδή οι σχέσει για σχέσεις πελατών και είχαν υποτιθεί σχετισμοί ότι ένα από τους λόγους πήγαινε αυτά, γιατί όλοι ψάχνουν το γιατί, τι γίνεται όσον αφορά αυτές τις ε, υποκλοπές των δεδομένων και ε, λέχθηκε ότι ένας από τους λόγους είναι ότι οι πληροφορίες περνούν από την υπηρεσία πληροφοριών στις διοικητικές αρχές. Και αυτό γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Και εδώ μας ενδιαφέρει εσείς πώς το βλέπετε από πλευράς δικηγόρου που δράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Κατά τη γνώμη μου σας γίνεται κάτι τέτοιο. Και αν ναι, πόσο αυτό παραβλάπτει το έργο εκείνων που δουλεύουν σε αυτό το περιβάλλον πώς επηρεάζει τα του ποινικού δικαίου. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός ε, αντίστασης του ΣΥΠΗΝ. Περισχυρισμών πρόκειται. Αλλά μας ενδιαφέρει να μας τα πείτε. Και θα σας πει η Σοφία Νιτφέλτ ε, τις δικές της ιδέες. Όλες μαζί τις ε, απαντήσεις, αν δεν σας πειράζει. Ναι, εντάξει, όλες μαζί. Θα μας πει τώρα η κυρία Μετφέλτ, κατόπιν ο κύριος Άλμπρουκ και κατόπιν θα λέτε λόγο εσείς κύριε Γκολ. Μερικές ερωτήσεις κι εγώ. Δεν είναι ε, νομική εμπειρογνωμών, αλλά νομίζω ότι στοχευμένη παρακολούθηση τον ακριφακούει κανείς ε, τις συζητήσεις δικηγόρου πελάτου είναι κάτι που επιτρέπεται με πολύ, σε πολύ πρεσμένες περιπτώσεις με δικαστική, ειδική δικαστική εντολή. Στοχευμένη παρακολούθηση σε μαζική κλίμακα είδαμε να έχουμε εδώ. Και αυτό που ε, προκύπτει είναι ότι οι δικές σας ανακοινώσεις είναι μέρος των παραλευμάτων, ε, για να το πω έτσι. Ως δικηγόρος θα λέγατε ότι αυτό είναι νόμιμο. Μπορεί κανείς να μηνύσει την κυβέρνηση, να μηνύσει τις μυστικές υπηρεσίες, διότι παραβιάζουν το δικό σας δικαίωμα, ακόμη και αν δεν το κάνουν ε, κατά πρόσωπο ή επίτηδες. Αν πάντως η δική σας ένωση θίγεται ε, παρεμπιπτόντος, γιατί δεν μπορώ να βρω τον κατάλληλο νομικό όρο, και εφόσον παραβιάζεται όχι ακριβώς ε, το επαγγελματικό απόρριτο, αλλά ισχύει εμπιστοσύνη μεταξύ δικηγόρου και πελάτου. Αυτό θα ίσχυε και για άλλα επαγγέλματα, φαντάζομαι. Του γιατρού, λόγω χάρη, και δικέ του επικοινωνίε κανονικά πρέπει να προστατεύονται και συμπεριλήφθησαν στην ε, μαζική παρακολούθηση και των δημοσιογράφων. Οι ε, γιατροί και δικηγόροι είναι σίγουρα διαφορετική κατηγορία από του δημοσιογράφου. Και αν οι συνομιλίες με τους πελάτες ήταν ένα παρακλάδι των παρανόμων πράξεων των μυστικών υπηρεσιών. Θα μπορούσε να, να γίνει κάτι γι' αυτό. Τι πιστεύετε. Και ακόμη με ενδιαφέρουν τρεις συστάσεις που ε, παρουσιάσατε. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο στο πώς θα γινόταν αυτό θεσμικός. Έχετε κάποια έτοιμη πρόταση. Έχετε προετοιμάσει Κάτι που θα μπορούσε να δώσει ιδέες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κ. Σόλμπρεχτ. Να συνεχίσω ακριβώς από αυτό που είπε η Σόφη. Για τις τρεις συστάσεις σας και εγώ θα ήθελα να ακολουθηθούν, αλλά οι πρώτες δύο ε, συνεπάγονται αλλαγή στη συνθήκη. Και η τρίτη θεωρήθηκε ανέφικτη από τον κύριο Γόλτερ από τα σχόλιά του στο προηγούμενο πάνελ. Μ' αρέσουν λοιπόν οι προτάσεις σας, αλλά πρέπει να πω ότι θα μου φαινόταν ε, πιο προβληματικό από ό,τι σε ένα σώθη. Δεν είναι απλώς ε, κάτι παράπλευρο. Στην περίπτωση Prism και την Tempora δεν τους νοιάζει πιανού τις επικοινωνίες αναλύουν ναι, και συγκεντρώνουν δεν έχει να κάνει με την ταυτότητα των ανθρώπων. Τους νοιάζει να αναλύσουν τα στοιχεία ολονών. Δεν τους νοιάζει ποιος είναι. Στο τέλος, που καταλήγουμε ότι με τα μέτρα παρακολουθήσεις που ισχύουν δεν υπάρχει πιθανότητα κατά την ε, διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων να διαλέξουμε υπέρ εμπιστευτικότητας μεταξύ συγκεκριμένων ε, συνομιλητών. Δεν υπάρχει πουθενά σκοπός συγκεκριμένος και εξειδικευμένος Δεν ξέρει κανεί σε ποια κατάσταση ανταποκρίνεται κάθε συνομιλία. Το θέμα είναι να μαζευτούν όλε. Αυτό μας οδηγεί βέβαια στην απεσιόδοξη στάση και εδώ πρέπει να μπει ένα απαγορευτικό όριο, διότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί δεν υπάρχει πλέον εμπιστευτικότητα μεταξύ δικηγόρου και πελάτου. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρόσφατα εγκρίθηκε οδηγία για το δικαίωμα πρόσβασης στους δικηγόρους, όπου ξεκάθαρα λέμε ότι η εμπιστευτικότητα στις σχέσεις δικηγόρου-πελάτου πρέπει να γίνεται σεβαστή από κάτι μέλη αλλά και αυτή η οδηγία έχει ένα παραθυράκι. Το παραθυράκι της εθνικής ασφάλειας. Οπότε το θέμα είναι ότι τι και να κάνουμε, πάντοτε θα σκοντάφτουμε σε αυτό το σκόπελο. Υπάρχει μια τεράστια μαύρη τρύπα. Εθνικής ασφάλειας, όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Ενώ τα κράτη-μέλη Μπορεί να μην έκαναν όλα όσα επιτρέπονται στο δικό του κράτο μέλο. Οπότε το θέμα είναι, πάτε πίσω στο δικό σα κράτο μέλο και το ρωτάτε εάν συμμορφώνεται με του κανόνε τη ECHR όταν ασχολείται με θέματα εθνική ασφάλεια. Νομίζω ότι οι αποφάσει τη ECHR και η ίδια ECHR αυτά που ισχύουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο με το αντίστοιχο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, θα πρέπει να δούμε ε, όλα αυτά θα μπορούσαν να ισχύουν και στις πολιτείες με το NSA, εάν θέλανε. Αλλά σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε. Και θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες τέλο πάντων. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε. Και στο προηγούμενο έγγραφο, αυτό που πρέπει να μα απασχολήσει ακριβώς είναι τι εννοούμε με την ηθική ασφάλεια και ποιε είναι οι εξαιρεσει όταν μιλάμε για την οδηγία και την πρόσβαση σε δικηγόρου και την εμπιστευτικότητα. τα μέτρα που εννοούμε καλύπτονται με μια περιοριστική ερμηνεία της ε, εθνικής ασφάλειας μέσω των συνθήκων. Κύριος Γκόλτσμιθ, μάλιστα για το πρώτο ερώτημα περί διαρροής μυστικών ε, που θα πάνε στις διοκτικές αρχές. Οπωσδήποτε δεν μας ικανοποιεί κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε, βλέπουμε το ζήτημα απόλυτα, έτσι όσον αφορά το επαγγελματικό απόρριτο τώρα με την ε, νομοθεσία περί ξεπλήματος χρήματος είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν υποψίες ε, οι δικηγόροι, στις διοκτικές αρχές και δεν μας ικανοποιεί αυτό καθόλου. Προσπαθούμε να το ανατρέψουμε. Οπότε, σε όποιο κράτο, κράτος μέλος και αν είναι κανείς, οι κανόνες διαφέρουν. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, εξαιρέσει, π.χ. αν η ζωή, είναι υποχρεωμένος κάποιος να αναφέρει κάποια πράγματα, αλλά κατά, είναι απόλυτο, κατά κανόνα είναι απόλυτος ο κανόνας. Και δεν θέλουμε βεβαίω ε, και τη δυνατότητα πρόσβασης των διοκτικών αρχών. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Το ερώτημα τώρα της κυρίας Ινετφέλντ για τις παρακολουθήσεις και το εάν είναι παράνομες ή όχι. Ε, αυτό εξαρτάται οπωσδήποτε το κάθε κράτος μέλος. Αυτή τη στιγμή ερευνάμε τις ε, δυνατότητες ε, των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση ε, στο απόρριτο. Είπα, όπως εμείς είμαστε κάθε, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις. Κάθε κράτος μέλος, μάλιστα, έχει διαφορετικές εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει γενική απάντηση αν είναι παράνομο ή όχι. Εξαρτάται από το Σύνταγμα. Ακόμα και το επαγγελματικό απόρριτο ε, διατυπώνεται διαφορετικά. Σε άλλες χώρες είναι στο Σύνταγμα, αλλού στον ποινικό κώδικα, αλλού είναι απλά ένας ε, κανόνας ο οποίος ε, εφαρμόζεται στα δικαστήρια. δικονομικά για τα αποδεικτικά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει εξαρτάται. Και βεβαίως υπάρχουν, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα άρθρα 6, 7, 8. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση εδώ πέρα μας βοηθάει πάρα πολύ και παρέχει μια γενική προστασία, αλλά στο εθνικό επίπεδο πριν πάει κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο το τι γίνεται. Τώρα το αν ισχύει για άλλους, ναι, το εάν τώρα είναι το ίδιο με τους δικηγόρους, κοιτάξτε, εγώ είδα μια δήλωση ε, προετοιμαζόμενος για να έρθω και είδα πως στους δικηγόρους, ε, οι δικηγόροι είναι οι μόνοι στους οποίους, για τους οποίους ισχύει ε, προστασία διανόμου του επαγγελματικού απορρίτου. Προφανώς δεν μπορώ να απαντήσω για όλα τα υπόλοιπα. Ε, τώρα, για το άλλο ερώτημα, είναι κάπως ε, ένα διπλό ερώτημα, δεν το είχα σκεφτεί. Θα μπορούσαμε ίσως ε, μέσω της δικής μας επιτροπής που έχει νομικούς να σκεφτούμε κάποιες προδιαγραφές. να σας βοηθήσει, ευχαριστώ. Ε, άκουσα αυτό το οποίο είπατε, πως δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, πως είναι άσκοπο. Ε, προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι άσκοπο. Χρησιμοποιούμε συχνά το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο αναπτύσσει επαγγελματικές πρωτεγραφές διατάξεις που τις χρησιμοποιούμε όταν απευθύνουμε επιστολέ στι κυβερνήσει και λέμε δεν συμμορφώνεστε με το ΧΙΨΙ ΜΕΓΑ, όταν υπάρχουν δικηγορικοί σύλλογοι του οποίου βοηθάμε να αναπτύξουν τέτοιε πρωτεγραφές, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα επιβολής, νομίζω πως οι προδιαγραφέ αυτές χρησιμεύουν και θα είναι και στο μέλλον χρήσιμε αν αλλάξουν ποτέ οι αρμοδιότητες. Οπότε ε, βοηθάνε όλα αυτά στο να αναπτυχθεί, αναπτυχθούν κάποιες, κάποια πρότυπα. Τέλος, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Άλμπρεχτ, όλα μαζεύονται και δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεση των δικηγόρων. Σε τεχνολογικό επίπεδο δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνολογικός, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πάντα είναι δυνατά και πρέπει να είναι δυνατόν εάν αναγνωριστεί το επαγγελματικό απόρριτο των ε, δικηγόρων και δεν ξέρω, αν, λέω εγώ διάφορα έτσι, αν βάλουν έναν ε, κώδικα ας πούμε, αν γράψουν κάτι να εξαιρέσουν τους δικηγόρους, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί τεχνολογικά να είναι εφικτό, αλλά ίσως να είναι κάπως δύσκολο. Ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις σας. Ο πρόεδρος ευχαριστούμε. Θέλει κανείς το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε. Και θα συνεχίσουμε στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα στις 9 Δεκεμβρίου. Στις 7.30 στο Στρασβούργο. Είναι εβδομάδα Λομελίας. Τι να κάνουμε, σε ποια αίθουσα δεν ξέρω. Συγγνώμη, συμπαθέτε μου. Θα μάθετε, θα υπάρξει ανακοίνωση. Ευχαριστούμε, γεια σας.